Uh, dear colleagues, Τι, να γελάσουμε όλοι, πείτε μας γιατί γελάτε. Ε, ε, ε, αναρωτιόμαστε πού έκανε διακοπές ο κύριος Σταυρακάκη. Σίγουρα όχι στις Βρυξέλλες γιατί έχει πολύ ωραία όψη. λένε, λένε ότι είναι στην πλάζ όλη την ώρα οι Έλληνε, αλλά δεν είναι αλήθεια, δουλεύουν σκληρά. Θα αρχίσουμε. Δεν θα έρθουν άλλοι. Και αυτό κάνει εντύπωση. Γιατί είναι η τελευταία έκθεση πριν από την τελευταία. Και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουν όλοι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, θα κάνουμε τα συνήθη, ό,τι κάνουμε τον τελευταίο χρόνο. Θα ακούσουμε από τους εισηγητές μια έκθεση πρόοδου αν θέλετε στις διαπραγματεύσεις για τους διάφορους κανονισμούς ενημερώνω ότι ε, ενώ υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να τύχουν επεξεργασίες λόγω της οριζόντιας φύσης των θεμάτων και θα αποφασιστούν στο γενικό κανονισμό, μιλάμε για αιτιολογικές σκέψεις, αλλά λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, τις εξαιρέσεις πρέπει να πω ότι οριστικοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και την εδαφική συνεργασία και για τους ομίλους, τον Ευρωπαϊκό Όμιλο. Θα υπάρξουν και άλλες ε, διορθώσεις όταν οριστικοποιηθεί ο Γενικός Κανονισμός. Αρχίζουμε με τον Γενικό Κανονισμό ε, και την Κωνσταντσε και μετά θα μιλήσουμε για το Ταμείο Συνοχής, γιατί ο Βίκτορ Μποστινάρου θα πρέπει να φύγει για το αεροδρόμιο νωρίτερα. Λάμπερ, Λάμπερ, μεγαλύτερη ομάδα πρώτα. Είμαστε ευτυχείς και η Κωνσταντζή και εγώ και οι Σχιώδης και εσείς οι πρόεδρος. Ε, είμαστε ικανοποιημένοι από τον τριμερή διάλογο, προσεγγίζουμε. Βέβαια πολλές φορές χρειάζεται πολύ υπομονή και δυναμικότητα και υπομονή. Την περασμένη φορά σας είπαμε ότι πολλά κεφάλαια ήταν ανοιχτά Υπήρχε όμως η επιθυμία να κλείσουν. Και εν προκειμένου έχουμε να πούμε καλά πράγματα για την Κομισιόν που μας βοήθησε και μας ε, ενθάρρυνε με κείμενα όταν χρειάζονταν να συγχαρούμε και το Συμβούλιο γιατί άλλαξαν το διαπραγματευτή και αυτό ήταν το καλύτερο που είχαν να κάνουν βέβαια γιατί ε, κάποιος ε, ε, διοικητικός μπορούσε να εξηγήσει αλλά δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί. Τώρα άλλαξε η ατμόσφαιρα και τα στρατόπεδα προσέγγισαν το ένα το άλλο. Και έχω την αίσθηση ότι και η Ιρλανδική Προεδρία ήθελε πολύ να συμβάλλει αποτελεσματικότερα από ότι στην αρχή του χρόνου. Πρόοδος λοιπόν, σημαντική. Δεύτερον, όπως είπατε, προετοιμαζόμαστε για τις ψηφοφορίες τον Ιούλιο και θα κάνουμε πιο λεπτομερή συζήτηση, αλλά η γενική άποψη είναι ότι όλα τα κεφάλαια άνοιξαν, αρκετά έκλεισαν και σε κάποια κεφάλαια υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμών σημείων που πρέπει και αυτά να οριστικοποιηθούν. Εμείς ε, έχουμε την ε, εντολή μας και αυτό θα μεταφραστεί και στον κατάλογο ψηφοφοριών που θα ετοιμάσουμε τον Ιούλιο. Αν δείτε όλα αυτά που συζητήσαμε, ε, το 90% των άρθρων έχουν ήδη τελειώσει, έχουμε συμφωνία. Να πω επίσης ότι είμαστε ευτυχείς διότι οι βασικοί κανονισμοί για το Ταμείο Συνοχής, το ΕΤΠΑ κλπ. προχωρούν. Και έχουμε ένα πακέτο κανονισμών έτσι που μπορούν να ψηφιστούν από την Επιτροπή μας. Υπ' αυτή την έννοια όλα βαίνουν καλώς, συμπλέουν. Και τονίζω ότι και εμείς στο γενικό κανονισμό θα στηριχθούμε όσο γίνεται περισσότερο στις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στους ε, πέντε διαφορετικούς βασικούς κανονισμούς. Αλλά εμείς έχουμε βεβαίως ε, σε τελευταία ανάλυση την ε, υποχρέωση τώρα να διαπραγματευτούμε για αυτά που μένουν να γίνουν, όπως για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα που δεν έχουν συμφωνηθεί. η Επιτροπή Απασχόλησης μιλάει για το 25% των διαρθωτικών και του Ταμείου Συνοχής που ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εντολή για τις διαπραγματεύσεις αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε όχι μόνο το 25% αλλά την απαραίτητη ευελιξία εκεί όπου γίνονται διαπραγματεύσεις. Και εκεί το Συμβούλιο έχει μια θέση ε, που δεν μπορούμε να τη δεχτούμε τώρα. Προσπαθούμε λοιπόν να ε, πάρουμε ό,τι μπορούμε από τις διαπραγματεύσεις. Τώρα, κάποια επιμέρους σημεία. Προφανώς η Κωνσταντζε θα επί τα υπόλοιπα ως συνήθως. Τώρα θα θίξουμε ακροθυγώς αυτά τα διακυβεύματα που υπάρχουν. Στην τέταρτη στήλη έχουμε ε, όλες τις λεπτομέρειες, όλες οι ομάδες. Θα αναφέρω ορισμένα μόνο από αυτά. Ένα από τα σημαντικά είναι η θεματική συγκέντρωση. Αυτή είναι η συνοχή 2.0 διαφορετικό από αυτό που κάναμε, γιατί είναι πολύ πιο έντονη η θεματική εστίαση και έτσι απαντάμε και στην κρίση και στο Ευρώπη 2020. Υπάρχουν μερικά που δεν τα έχουμε συμφωνήσει. Ευτυχώς ε, συμφωνήσαμε επί των περισσότερων από τους 11 στόχους στον έκτο στόχο θέλουμε προστασία του περιβάλλοντος, λέει διατήρηση. Θέλουμε να προσθεθεί η προστασία. Αυτό είναι στα πλαίσια της εντολής μας. Επίσης συζητήσαμε για τα δίκτυα και τις υποδομές ε, όπου συζητήσαμε για τα εμπόδια ε, τους κρίκους που λείπουν, πρέπει εδώ να ληφθούν υπόψη, η επιθυμία του ΔΕΚΑ επίσης δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με την επακριβή διατύπωση που θα, μιλά, θα αναφέρεται στους παλαιούς εμπλεκομένους. Αυτά μπορούν να προχωρήσουν. Και σας μίλησα τώρα τους, για τους θεματικούς στόχους που ευθυγραμμίζονται με αυτά που συμφωνήσαμε για το ΕΤΠΑ και το Κοινωνικό Ταμείο. Για το Κοινωνικό Ταμείο δεν ε, έχουμε συμφωνήσει και μάλιστα αυτό θα είναι ένα θέμα που θα αναδειχθεί αργότερα στη συζήτηση στην Ολομέλεια γιατί το Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει στόχους που και πρέπει να βρούμε κάποια μέσα τα οποία στο εσωτερικό της κάθε χώρας θα αποτελέσουν μια προσέγγιση ε, με προσανατολισμένη στην ζήτηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πόλεων και των περιφερειών. Ε, σημαντικό είναι να εξακολουθήσει να υπάρχει ευελιξία γιατί και του τριμερείς διαλόγους με την Κομισιόν και το Συμβούλιο σε υψηλό επίπεδο ε, είχαμε κάποιες διευκρινήσεις και με τον Επίτροπο Άντορ και με τον Επίτροπο Χάν και οι δύο υπέβαλαν προτάσεις και τους ζητήσαμε να υπολογίσουν πάλι τα αποτελέσματα που θα έχουν οι προτάσεις τους και να καταλήξουν σε ένα σύστημα που θα ανταμείβεται η ευελιξία. Για την εδαφική ανάπτυξη, σημαντικό θέμα, ε, υπάρχει συμφωνία. Ε, βρήκαμε πιο πολύ, εξασφαλίσαμε πιο πολύ υποστήριξη για την ανάπτυξη που θα καθοδηγείται από τις τοπικές κοινότητες ε, με την υποστήριξη διαφόρων ταμείων και εκεί ε, φροντίσαμε να υπάρχει ευελιξία. Έχει κλείσει αυτό το κομμάτι και υπάρχει δυνατότητα να γίνει χρηματοδότηση και από το ΕΤΠΑ και από το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Κάτι που σας είπαμε την περασμένη φορά επίσης για το κοινό πλαίσιο στρατηγικής. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος εργασίας για το Κοινοβούλιο εδώ. Θυμάστε που στο Κοινοβούλιο είχαμε ετοιμάσει ένα παράρτημα το οποίο τώρα έχει, έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο ως σημαντικό μέσο ώστε να γίνεται συντονισμός και συνδυασμός των ταμείων λαμβάνοντα υπόψη και το Horizon ή άλλα ταμεία εκτός από το αυτά των πέντε κανονισμών ή αυτά που λειτουργούν στο περιβαλλοντικό τομέα και σε στην πράξη διευκρινίζεται ο τρόπος χρήσης των ταμείων, τι είναι επιλέξιμο, ποια θα είναι η διαδικασία, όλα αυτά είναι σημαντικά και τα δέχτηκαν στο Συμβούλιο, στην Κορεπέρ, παρουσίασαν κάποια τεχνικά ζητήματα που πρέπει να ε, διασφαλιστούν και βλέπουμε τέλος ότι με την συνομοθετική δράση του Κοινοβουλίου μπορούμε να ασκήσουμε μεγάλη επιρροή. Ε, αφιερώσαμε χρόνο για αυτές τις διαπραγματεύσεις και βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα ότι τα εθνικά κράτη είναι τόσο διασπασμένα και ακόμα δηλαδή ε, υπάρχουν αρνητικά σημεία στη συζήτηση, υπάρχει δηλαδή, ε, υπάρχουν οι φίλοι της συνοχής, ε, οι φίλοι της καλύτερης χρήσης των δαπανών που δεν ήταν πρόθυμοι να ρίξουν γέφυρες μεταξύ των ταμείων και εκεί παρενέβη το Κοινοβούλιο και έκανε πολύ καλή δουλειά που οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου συστήματος πολυχρηματοδότησης παρά την ε, χωριστή μόνο χρηματοδότηση του παρελθόντος. Ε, γιατί ε, δημοσιονομική διαχείριση. Έχουμε κάποια θέματα για τις πληρωμές, τις διορθώσεις, τους τελικούς δικαιούχους. Εδώ υπάρχουν πολλά άρθρα τα οποία συμφωνήσαμε όμως. Τα οικονομικά θέματα ε, είναι ακόμα ανοιχτά σε μεγάλο βαθμό δίχτυα ασφαλείας ε, για τις περιφέρειες 2007-2013 ε, νησιωτικές περιοχές, το ΣΕΦ, αυτό το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, καθορισμός του ποσοστού συγκριματοδότησης, πληρωμές, ε, η προχρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική και εδώ ε, μένουμε στη θέση μας. Ε, τα χρηματοδοτικά μέσα τώρα ε, συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν πολλά στοιχεία, κάποιες προσωρινές διατάξεις, ε, ένα θέμα παραμένει μόνο ανοιχτό εκεί. Ακόμα την επόμενη εβδομάδα, ε, την επόμενη εβδομάδα δεν πρέπει να ρυθμίσουμε τα εκρεμή που είναι πια όρημα φρούτα όμως για να συμφωνήσει το Συμβούλιο. Συνήθως η συνεισφορά της Κωνσταντσε ε, έχει, έχει μια ιδιαιτερότητα γιατί όλο άνδρες είναι εκεί και δεν μπορώ καμιά φορά να τους πείσω και μετά βγαίνει από τα χείλη της Κωνσταντσε η μαγική πρόταση και τους ποιήθη. Ε, για εξήγησε στα μέλη πώς θα καταφέρνεις. Η Κωνσταντσε ξέρει ότι εγώ ε, κάνω κουμάντο εδώ, δεν θα μιλήσει αν δεν της δώσω το λόγο. Και δεν υπάρχουν πια τόσα πολλά όρημα φρούτα, ε, θα είναι δύσκολα και για την Κωνσταντσε ναι, κανείς δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, να προσθέσω και εγώ μερικά για ότι έχουμε τελειώσει τώρα, για στατιστικούς λόγους. Κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει στα πλαίσια των ε, τριμερών διαλόγων. Στους τελευταίους τριμερείς μπορέσαμε να επιλύσουμε ορισμένα προβλήματα, ορισμένα ζητήματα με την Προεδρία. Ήθελα να πω το ίδιο που είπε και ο Λάμπερτ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους διαπραγματευτές, τη γραμματεία, την Πρόεδρο. Είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε συσπηρωθεί σε τόσο ε, δύσκολους ε, καιρούς και πολλές φορές ε, δεν είναι καθόλου εύκολο να συνεργαστούμε με την Ιρλανδική Προεδρή. Όμως, χτες κλείσαμε τρία ανοιχτά μπλοκ, κεφάλαια. Δηλαδή μετά από τρεις τριμερείς παρουσιάσαμε στην Προεδρία ένα πακέτο για διαπραγμάτευση και χτες ε, δώσαμε τελική μορφή στο πακέτο μέχρι την ε, ψηφοφορία στην Επίτροπη. Για αυτά τα τρία μπλοκ θα ήθελα να σας ε, μιλήσω. Ως προς την ε, εκλογιμότητα, καταρχήν, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να την διασφαλίσουμε στη διαδικασία απλοποίησης χωρίς ε, να βγάλουμε τις ρήτρε διασφάλισης που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ζήτησε κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο και θα διευθετηθεί. Αυτά στα οποία αναφέρομαι είναι τα πιο δύσκολα σημεία Διαφορετικά παραμένουμε στην εντολή μας με την Κομισιόν. Ήταν δηλαδή εύκολο να φτάσουμε σε συμφωνία σε πολλά επιμέρους σημεία, αλλά τα τελευταία άρθρα στις τελευταίες παραγράφους ήταν δύσκολα και ήταν χρονοβόρα η διαδικασία συμφωνίας. Στο άρθρο 55.6 υπάρχουν ε, διαφορετικά φορές ε, σε σχέση με την επιλογή, την επιλεξιμότητα των ε, δαπανών και φτάσαμε στη συμφωνία με το Συμβούλιο. Στο 58.1β αποφασίσαμε για ένα καταποκοπήν πόσο για, το, για τις δαπάνες προσωπικού, κάτι το οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις, ε, θα βοηθήσει τις, διαδικασίες για το διοικητικό, ε, οι διοικητικές δαπάνες. Άρθρο 58.2 ώρες εργασίας για το προσωπικό εδώ είχαμε μία μακροχρόνια συζήτηση, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα εθνικά συστήματα, τους εθνικούς νόμους για αυτή την καταμέτρηση. Δεν καταλάβαμε γιατί η Προεδρία ήθελε να μπουν αριθμητικά στοιχεία σε αυτή την παράγραφο και τέλος συμφωνήσαμε με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο 1720 ώρες δηλαδή. Ακούγεται απλό, όμως ε, αυτό σημαίνει ότι θα γίνει υπερχρηματοδότηση σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτή θα είναι η φυσική συνέχεια. Και εμείς δεχτήκαμε το μέσο ευρωπαϊκό όρο για να φτάσουμε σε συμβιβασμό. Στο άρθρο 59.3β ο κύριος Ζήμαν δεν είναι παρόν, δυστυχώς, για να μας το επεξηγήσει υπήρχε διαφορετική άποψη ενός μέλους. δηλαδή να υποστηρίξουμε εκείνους οι οποίοι είναι υπέρ του brownfield και όχι του greenfield. Ε, ε, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν παλιές εγκαταστάσεις και όχι νέες και μιλάμε για 15% δηλαδή για ε, συγκεκριμένα σημεία βιομηχανικής χρήσης και κρίναμε ότι θα πρέπει να δοθεί συνέχεια για την χρήση τους. Στο 59.3 γάμα σε σχέση με το ΦΠΑ που δεν ανακτάται, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία, είδαμε ε, ότι επιμείναμε και κερδίσαμε. Στο άρθρο 61 παράγραφος 1α, καινούρια 1α, πρόκειται για ένα άρθρο για την επανακατανο... μάλλον για την επαναγκατάσταση των επιχειρήσεων και όπως ξέρετε αυτό είναι ένα θέμα πολιτικής υφής Μετά από τις κρατικές ενισχύσεις η Προεδρία δέχτηκε η επανεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε μία δεκαετία να επιτραπεί. Και σε αυτή την περίπτωση θα επανακτηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ισχύει για τις ΜΜΕ, αλλά όπως ξέρετε είναι μία μακροχρόνια θέση μας και ε, επιτύχαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε την τελική έκβαση, η πενταετία είναι ο βασικός κανόνας και η τριετία για τις ΜΜΕ. Αυτός είναι, αυτή είναι η τρέχουσα πρακτική και 10 χρόνια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 114, είχαμε μακρά συζήτηση για την ε, αναλογικότητα και έλεγχο των προγραμμάτων και φτάσαμε σε μία συμφωνία όπου ε, προβάλλεται αύξηση των κονδυλίων με ε, ελέγχους από το Συμβούλιο, κατόπιν ελέγχων από το Συμβούλιο. Είναι όμως εξισορροπημένη θέση και προς τις δύο κατευθύνσεις και ευχαριστούμε την Επιτροπή που μας ναι. βοήθησε σε αυτό το σημείο. Ναι. Το επόμενο μπλοκ είναι ο έλεγχος και η αποτίμηση και εδώ προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε το ρόλο των επιτροπών εποπτείας. Άρα τα πιο δύσκολα άρθρα ήταν το 42 παράγραφος 1 όπου θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία έτσι ώστε οι ε, επιτροπές ελέγχου να αποφασίσουν κατά πόσο υπάρχει δικαίωμα ψήφου και δυνατότητα ε, ψηφοφορίας ε, στις επιτροπές αυτές. Υπήρχε κόκκινη γραμμή από τα κράτη-μέλη αρχικά και γι' αυτό η επιτυχία μας ήταν ακόμα μεγαλύτερη ιδιαίτερα ε, για τις μη κυβερνητικέ και τους κοινωνικούς εταίρους. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Στο άρθρο 43.3 οι επιτροπές ελέγχου μπορούν να γνωμοδοτήσουν όταν τροποποιούνται τα προγράμματα. Στο 44.8 μιλάμε για την πλήρη ετήσια εφαρμογή ε, του προγράμματος σε σχέση με στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται για τους πολίτες προς τα έξω δηλαδή, η Προεδρία είχε ταχθεί κατά της περαιτέρω διαφάνειας και πληροφοριών προς το κοινό. Τελικά ε, επιτύχαμε και πάλι, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η διαπραγμάτευση. Στο άρθρο 101 παράγραφος 3 προσθέσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα για ε, αμαία και προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και για την απασχόληση των νέων, για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Αυτό ήταν ένα πολύ ε, έντονο πολιτικό θέμα για μας. Στο 102 μπορούμε να αυξήσουμε τη διαβίβαση των στοιχείων προς την Κομισιόν από δύο σε τρεις φορές ετησίως. Αυτό είναι συμβιβασμός. Αν παρακολουθήσατε τις ε, διαπραγματεύσεις για τον ε, διορθωτικό προϋπολισμό και τη νέα διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι έχουν τα σωστά αριθμητικά στοιχεία και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό η Επιτροπή και, η και το Κοινοβούλιο ζητούν μεγαλύτερο προϋπολογισμό από πλευράς πληρωμών. Τώρα έχουμε μια καλύτερη βάση για λήψη αποφάσεων και τα κράτη-μέλη μπορούν ε, να μας πούν, ε, μπορούν να μας αποστείλουν τα στοιχεία τον Ιανουάριο, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Τρεις φορές δηλαδή το χρόνο. Γι' αυτό ήταν για μας ε, μεγάλη επιτυχία και στη συνέχεια είχαμε μία τροπολογία από το Κοινοβούλιο για, το ένα, για ένα νέο άρθρο 48 Β εξάντε αξιολόγηση των ε, μέτρων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου ε, για τους δικαιούχους και αυτό είναι πολύ θετικό. Διαπραγματευτήκαμε αυτό το νέο άρθρο γιατί όλοι βεβαίως αναφέρουμε και λέμε ότι θέλουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία αλλά άλλο να λέμε, άλλο να κάνουμε. Όταν πρέπει να αξιολογήσουμε τα μέτρα είναι πολύ πιο δύσκολο να πούμε ότι θέλαμε αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν να μειώσουν το γραφειοκρατικό φόρτο. Στο 101α δίνουμε περισσότερο χρόνο στα κράτη-μέλη για, την, για τις εκθέσεις πρόοδου και εφαρμογής. Βεβαίως κάθε διαπραγμάτευση αποτελεί συμβιβασμό και γι' αυτό έπρεπε να δώσουμε και κάτι στην Προεδρία. Ε, πληροφορία, πληροφόρηση, επικοινωνία και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν το επόμενο μπλοκ αυτό το μπλοκ είναι σημαντικό και για λόγους διαφάνειας, αλλά και για να προωθήσουμε την πολιτική και ανταλλαγή ε, στοιχείων μεταξύ εντολέων και δικαιούχων. Στο άρθρο 105β μιλήσαμε για μία ενιαία ιστοσελίδα που θα δίνει πληροφορίες για ε, επιχειρησιακά σχέδια, καθώς και την προθεσμία, τις προθεσμίες με βάση μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Αυτό είναι πολύ θετικό για τη μελλοντική μας πολιτική. Στο 105.2 μιλήσαμε για διαφάνεια. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να δώσουν μια συγκεφαλαίωση των προγραμμάτων, των ε, προγραμμάτων αυτών που θα ενημερώνονται κάθε έξι μήνες. Στο παράρτημα 6.2ε αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να δημοσιεύσουμε ορισμένα παραδείγματα ε, δράσης, ε, ε, δηλαδή στην ιστοσελίδα στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ιρλανδοί επειδή μιλούν αγγλικά δεν θέλουν να λάβουν υπόψη μια οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Για εκείνους είναι εύκολο για την Εσθονία, για την ε, Ουγγαρία ή την Ελλάδα είναι κάτι το διαφορετικό. Και για την Ελλάδα μόνο μερικοί, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευρέως κατανοητά αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό θέλαμε να γίνει μετάφραση τουλάχιστον ως προσωρισμένα προγράμματα και συμφωνήσαμε. Στο παράρτημα 6, παράγραφος 221β, αποφασίσαμε εάν υπάρξει συγχρηματοδότηση από πολλά ταμεία, τότε να δημοσιοποιηθούν τα μέτρα σε σχέση με κάθε ταμείο χωριστά. Να γίνει αυτό ή να μιλήσουμε μόνο στα, για τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων. Η Προεδρία δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει αυτό το θέμα και στο παράδειγμα στο άρθρο 3β μιλήσαμε για την διαχειριστική αρχή η οποία θα πρέπει να δώσει τις πληροφορίες ε, στα γραφεία πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δυστυχώς ε, δεν μπορέσαμε να εισαγάγουμε όλα τα, όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η συμφωνία και συμμετέχουν και τα γραφεία πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επειδή θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να προβάλλουμε μια άλλη στρατηγική διαπραγματεύσεις. Πρότεινα ένα σύνολο τεσσάρων μπλοκ για να συμφωνήσουμε, διότι πολλές φορές είναι εύκολο να φτάσουμε σε συμβιβασμό εάν ε, υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες από αυτές του ενός ε, μπλοκ, γιατί σε κάθε μπλοκ υπάρχουν 6 με 8 σημεία τα οποία δεν έχουν συμφωνηθεί. Αυτό είναι μέρος της στρατηγικής της Προεδρίας. Υπάρχουν και προτάσεις συμβιβασμού, επιτάπητος, αλλά θέλουμε να έχουμε αυτό το, αυτή τη δυνατότητα ε, διαπραγμάτευσης. Μιλάμε για έλεγχο, διαχείριση, ε, προγράμματα που οδηγούν σε ε, υψηλές προσόδους και ούτω καθεξής. Θα προσπαθήσουμε στον επόμενο τριμερή να τα προωθήσουμε αυτά. Όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα εισαγάγουμε στην έκθεσή μας που θα ψηφίσουμε στις αρχές Ιουλίου. θα είναι συμβιβασμοί έτσι ώστε τον Ιούλιο να προωθήσουμε τριμερείς διαλόγους για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και θα μπορέσουμε να κλείσουμε και άλλες ενότητες, άλλα μπλοκ Ελπίζω να μας υποστηρίξετε για να κλείσουμε τις τέσσερις αυτές ενότητες με πολλαπλά σημεία και να φτάσουμε και σε συμβιβασμό στα δυσχερή εκρεμή σημεία. Σας ευχαριστώ όλους που μας υποστηρίξατε και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κατά τον επόμενο τριμερή. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας πω ότι ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διευθυνσής για τις Περιφερειακές Υποθέσεις τι να σας πω, είσαστε ο αρχιδιαπραγματευτής της Κομισιόν, θα το έλεγα, αλλά δεν διαπραγματεύεται η Κομισιόν, έτσι. Ε, και όμως πάντοτε έρχεται να μας δώσει την βοήθειά της. Οπότε, αν θέλετε, και αν συμφωνεί και η Κωνσταντζα μπορούμε να έχουμε συζήτηση, ερώτα απαντήσει τέλο πάντων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει κάποιο το λόγο. Απίστευτο. Αλλά πολύ καλό. Μπλάσο. Μπλάσα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας πω πόσο, πόσο αξίζουν συγχαρητήρια οι διαπραγματευτές μας και εγώ ίδιος έχω παραστεί σε μια σειρά από τριμερείς διαλόγους και όντως ε, όφυλαν όλοι να δουλέψουν σκληρά και καμιά φορά φτάσαμε τα μεσάνυχτα και οπότε δεν μπορώ παρά να δώσω συγχαρητήρια αλλά και να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, ε, πάντοτε είχαν στάσει πάρα πολύ επικοδομητικοί, είχαν πολύ καλή συνεργασία. Όμως, όσο αυτό το κεφάλαιο τώρα, ήταν θέμα της θεματικής συγκέντρωσης, γιατί ήταν θέμα επίσης προετοιμασίας και συμφωνίας για την συνεργασία ούτω ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα λειτουργικά προγράμματα, του θεματικού στόχους ε, που δεν υπήρχαν πάντα ή να υπάρχει κάποιο είδου κατανομή των πόρων. Όλα αυτά ήταν ένα έργο που πρέπει να επιτελεστεί και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, που συμμετείχαν και η προετοιμασία προς τούτο. Στο, αλλά σχόλια λέει ο Πρόεδρος Λαμπέρ εμφανίστε εδώ. Και εγώ και η Κωνσταντζα Ήθελαμε πρώτα να ξέρουμε από πού ξεκινάμε, πού στηριζόμαστε για αυτές τις διαπραγματεύσεις και πάνω το θέμα αυτό είναι μια καυτή πατάτα. Ε, ρίξτε μια ματιά στο τι γίνεται. Είναι υπέροχο αυτό το οποίο συμβαίνει και συμβαίνει. Το, το ότι θα πρέπει τελικά να μήψουμε, να επενέσουμε τα καλύτερα προγράμματα. Είναι, μπαίνουν στην άκρη τα χρήματα και μετά αποδίδονται. Οπότε και αυτό ήταν ένα θέμα στις διαπραγματεύσεις η καυτή πατάτα που δεν αρέσει. Το θέμα είναι πώς αυτό μπορεί να το διαπραγματευτεί, πώς αυτό να το χειριστεί τραπέζες, γιατί είναι σαφές ότι αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε στα πλαίσια της συζήτησης για το 5% για το πολιετές πλαίσιο. Άρα θα πρέπει κανείς να είναι ικανοποιημένος ποιος. Ο Κάμερον, όχι ο Κάμερον. Εμείς. Μια που κάτι αποσπάσαμε. Το άλλο είναι η μακροοικονομική ε, εξάρτηση. And to see how to bring them because to an end and uh, αυτή η αιρεσιμότητα τέλος πάντων για να δούμε πώς θα συμπληρωθεί αυτή η δέσμη μέτρων. Οπότε έτσι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή φέτος κάποια στιγμή. Άρα δύο είναι οι καυτές πατάτες. Οπότε επίσημα ή Επίσημα, Αν έχετε κάποια συμβουλή να μου τη δώσετε. If there no, more, uh, yes, uh, who was first? Uh, Jan Albrecht, and then. Jan Ευχαριστώ. Έχω τις εξής τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα, όπως και ο Βλάσακ, θέλω να σας πω ότι και εμείς περιμένουμε να γίνει θεματική συγκέντρωση του Κοινωνικού Ταμείου. Οπότε πια να έχουμε μια αποδόμηση ούτως υπήν του όλου συστήματος. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε επιγόντως Πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις ξανανοίγουν και να δούμε τελικά ποιο πρότυπο θα γίνει αποδεκτό. έχοντας όλη επίγνωση των συνεπειών της συγκέντρωσης. Υπάρχουν κάποια σενάρια, ελπίζω δεν ελθεύουν και η θεωρητική πιθανότητα αλλαγής των θεματικών στόχων. Αν ε, κάποιος θέλει να αλλάξει τα ονόματα αυτών των στόχων, τότε θα είμαστε παγιδευμένοι. Τώρα το τελευταίο στοιχείο είναι αυτό το οποίο πριν από λίγο ο Λάμπερτ. Το θέμα του, της, ε, του αποθεματικού της επίδοσης των επιδομάτων αφορά το 7% που όπως έχει ρυθμιστεί. Αλλά αυτό είναι η προϋπόθεση ούτως ώστε οι πληρωμές να είναι στο επίπεδο του 1908 και το συν 3%. Οπότε το σύστημα όλο αυτό, όπως το έχει προτείνει το Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να ζητηθεί δεν θα στέκει. Ή μάλλον θα στέκει, θα είναι εφικτό. Αλλά θα γίνει τόσο δύσκολη η εφαρμογή των πολιτικών αυτών που κανείς δεν θα μπορεί να προχωρήσει. Και έτσι θα έχουμε οικονομία αστείο. Βέβαια αυτό ίσως χρειάζεται να γίνει έτσι μια που υπάρχουν τόσο λίγα χρήματα. Από πλευρά συστημικής τώρα έχω κάποιες ε, επιφυλάξεις πάντως για τις πληρωμές εγώ διστάζω να έχω αντίρρηση. Τελικά το ζήτημα είναι αν όλα αυτά είναι εφικτά. Αυτό και να δούμε αν αυτό που αποφάσισαν οι Υπουργοί Οικονομικών θα είναι ρεαλιστικό. Μιλάμε για το 2021, 2022, 2023, αυτό το 7%. Δηλαδή έτσι μετέθεσαν το πρόβλημα πιο αργά. Ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι. Ο Λάμπερτ μίλησε για τα κεντρικά προβλήματα και καταλαβαίνω τους συναδέλφους στους άλλους τριμερείς διαλόγους. Προσθέτω και τον τριμερή για το ΕΚΤ που θα πρέπει να εξετάσει την ε, θεματική εστίαση, η συγκέντρωση. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που εξαρτάται από αυτήν. Ε, τα, τα ανοίξαμε έγκαιρα με την επικυπριακή προεδρία κλείσαμε κάποια... Είχαμε αρχίσει διαπραγματεύσεις ε, με κάποια, για κάποια κεφάλαια, όπως για τον προγραμματισμό, που, τώρα, που μετά όμως μπήκε στο ντουλάπι και δεν ξαναβγήκε. Ε, ήταν, οι ε, Ιρλανδοί έβαλαν κάποιους, κάποιους όρους εκ των προτέρων που δεν τους κατάλαβα απόλυτα. Ε, ε, είδα ότι μπλοκαρίστηκαν όμως κάποια θέματα. 40 τριμερείς διάλογοι βέβαια έγιναν, υπήρχε δυνατότητα να διαπραγματευτούμε οι έμπειροι δηλαδή ξέρουν ότι εκεί δεν είχαμε πρόβλημα. Ε, 16 Μαΐου θέλαμε την τελευταία φάση, μετά είχαμε κανονίσει ο καθένα τις δουλειές του και τώρα ε, βλέπουμε ότι τα ανοιχτά θέματα είναι περισσότερα. Κάποια είναι κεντρική σημασίας, ε, τρία θεωρώ κεντρικά, τέσσερα μάλλον, που μάλλον θα μας απασχολήσουν μέχρι το τέλος και, γιατί επηρεάζουν και τις, τους άλλους κανονισμούς. Ε, είναι το μερίδιο του ΕΚΤ, προσπαθούμε εδώ να ε, επιτελέσουμε πρόοδο, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί διαπραγματεύεται επί άλλης βάσεως το Συμβούλιο και δεν συμφωνούμε ούτε επί της διαπραγματευτικής βάσης. ή εκ των προτέρων ερεσιμότητες για τις οριζόντιες πολιτικές είναι το δεύτερο σημείο. Επίσης αυτό το αποθεματικό επιδόσεων, το performance reserve είναι ένα σημαντικό θέμα και το πιο σκληρό είναι η μακροαιρεσιμότητα. μακροκοντισιονάλιτη, μακροοικονομική. Τέσσερα λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο δεν το έχουμε ανοίξει και είναι σαφές γιατί, θα είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί αυτά τα τέσσερα κεφάλαια να σέρνονται μέχρι το τέλος. Ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε για, τα, για τους τίτλους των κεφαλαίων. Ε, εδώ έχουμε κάνει καλή δουλειά. Και δεν θέλουμε να αφήσουμε το θέμα. Κάθε διαπραγμάτευση άλλωστε ε, είναι, στοιχίζει ένα κομμάτι από τη δική μας την εντολή, το ξέρουν οι διαπραγματευτές. Δεν θέλουμε αυτά που κουραστήκαμε να πετύχουμε να τα χάσουμε, όμως Έχουμε ε, τίτλους ε, θεματικής συγκέντρωσης στο άρθρο 9 που συζητήθηκαν σε πολλούς τριμερείς διαλόγους και χρειάζεται κάποια ε, επιδεξιότητα από την πλευρά μας ούτως ώστε να υποβάλουμε μια γενικότερη συνολική πρόταση στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να ζυγίσουμε τα Δούνε και Λαβίν και να δούμε αν στις διαπραγματεύσεις θα βρούμε μια λύση. Ε, με την Κομισιόν συνεργαζόμεθα καλά. Ε, ελπίζουμε ότι θα συμπαρασταθεί. Δεν νομίζω ότι στο άρθρο 9 είναι η τίτλη ε, το πρόβλημα. Το βασικό είναι το θέμα της συγκέντρωσης, θεματική συγκέντρωση εστίαση, thematic concentration. Αυτό δεν βλέπω να λύνεται εύκολα. Για Αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να το πούμε. Ιδιαίτερα επειδή υπάρχει αυτή η βασική στάση του Συμβουλίου ότι ε, δεν θέλει να διαπραγματευτεί. Και η Ιρλανδική Προεδρία δεν μας έπεισε για το αντίθετο, ότι δηλαδή αλλάζει λίγο, είναι προετοιμασμένη να, κάνει, να αποκλείσει, να μπλοκάρει πράγματα, όχι να, να διαπραγματευτεί. Και το βλέπουμε αυτό ε, και από πριν. Όταν ρωτάμε δηλαδή ποια είναι η πρότασή σας στις διαπραγματεύσεις, βλέπουμε ότι σιωπούν και αναβάλλεται το κεφάλαιο για την επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα είναι γνωστό ότι πια ε, υπάρχει αυτή η ε, δυσαρέσκεια. Γιατί πολλές φορές με ρωτάνε γιατί ε, δεν τελειώνουμε δεν έρχεσαι, πολλές φορές μου λένε και από την εκλογική μου περιφέρεια, δεν έρχεσαι. Μα οι τριμερεί διάλογοι, μα μας λε ότι είσαι στου τριμερεί διαλόγους, αλλά δεν τελειώνεται ποτέ. Πάντως ε, πρέπει ε, δημοσία να καλέσουμε και την Ολλανδική Προεδρία να κρατήσει τα προσχήματα, να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, γιατί αυτό είναι και ε, ένα τεκμήριο, αν θέλετε, της επιτυχίας της, στην Προεδρία. Δεν μου φαίνεται να θέλει άλλος να μιλήσει. Ο Βίκτορ, όχι. Α, η Κωνσταντσε μόνο. Μάλιστα. Μια σύντομη διευκρίνηση ε, μετά από αυτά που είπε και η Ελίζαμπεθ και ο Λάμπερτ πριν για το ΕΚΤ. Θέλω να κλείσει το θέμα εμείς ε, κάναμε τις προτάσεις μας και στα πλαίσια της εντολής μας η πρότασή μας ήταν έξυπνη για να εξασφαλίσουμε ευελιξία για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες χωρίς να χάνουμε από τα μάτια μας το στόχο μας. Αλλά από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο δεν θέλει καθόλου να παρεκκλίνει. Τώρα, ε, μετά από τα τέσσερα σημεία που ανέφερες εσύ, αν τα δούμε τα τέσσερα σημεία ε, μαζί, Ελίζαμπεθ, θα έλεγα ότι πέρα από πολιτικές παρατάξεις και από επιτροπές, ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί αν μπορούμε να παραμείνουμε στην ε, απόρριψη του performance reserve. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε που και για μας ανοίγουν κάποια περιθώρια. Μπορεί να μην είναι μεγάλα, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Γιατί όλους μας ενδιαφέρει μια συμβιβαστική λύση. Ας αρχίσουμε λοιπόν στο ένα ή στο άλλο σημείο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πού μπορούμε να κάνουμε υποχωρήσεις. Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι θα παραμείνουμε στην εντολή που έχουμε αναλάβει. Εκεί δεν τίθεται θέμα. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να περιχαρακωθούμε και να κάνουμε σαν να μην υπάρχει η πραγματική, ο πραγματικός κόσμος, η πραγματικότητα γύρω μας. Σκεφτείτε το. Να το έχετε στο μυαλό σας. Και καλό είναι να δώσουμε αν υπάρχουν και ε, κάποιες ε, σοφές οδηγίες ε, για το τι μελγενέστε στα περαιτέρω. Pierce? No. What are you saying? I, Joachim. Yeah. If you just do it like this, I can see it better. But if you just do it here, I don't see. Danke, Frau Vorsitzende. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς τους ε, συναδέλφους που είναι στη διαπραγματευτική ομάδα. Και πραγματικά σας βγάζω το καπέλο. 40 τριμερείς διάλογοι ε, αυτό στοιχίζει σε χρόνο, σε νεύρα, σε ποιότητα ζωής. Αλλά τι λέτε, πόσο θα συνεχίσουν όλα αυτά, για πόσο καιρό θα συνεχίσει αυτή η ιστορία. Ε, η Ιρλανδική Προεδρία πολλές φορές επικρίνεται. Εγώ μπορώ να πω ότι οι Ιρλανδοί με τους οποίους διαπραγματεύτηκα στα δικά μου θέματα ε, στα πλαίσια της γενικής οδηγίας ε, αυτό ε, εγώ είχα ένα ίσον θέμα αλλά είδα μεγάλη προθυμία αλλά οι καημένοι συνάδελφοι τι να κάνουν άνδρες ήταν ε, πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλους τους, και, το, 27. Και μετά την απόφαση το Φεβρουάριο το Συμβούλιο δεν ε, μετακινήθηκε γραμμή. Ε, μιλούν μόνο για τις θέσεις τους στα πλαίσια για το πολιετές δημοσιονομικό. Και τώρα ε, πολλοί απευθύνουν εκκλήσεις στις κυβερνήσεις ούτως ώστε να ε, γίνει, για να γίνουν κάποια βήματα. Άμα δεν φτάσουν αυτά μέχρι την Προεδρία όμως, και η καλύτερη Προεδρία να είναι, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Δεν έχει περιθώριο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ας σκεφτούμε κι εμείς πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Η πολιτική, η πολιτική συνοχή έχει το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού και στο Συμβούλιο, στο πολιτικό επίπεδο, ε, οι διαπραγματεύσει γίνονται από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για τα θέματα. α πούμε, Υπουργείο Εξωτερικών στη Γερμανία, συνάδελφοι από εκεί. Αυτοί δεν έχουν σχέση με διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχή, δεν τα ξέρουν καλά τα θέματα. Άρα εδώ έχουμε ένα διαρθρωτικό σφάλμα. Και το ερώτημα είναι αν τα κράτη-μέλη στην πλειονότητά τους ενδιαφέρονται να πετύχει συζήτηση. Θυμάστε τη συζήτηση πριν από δύο-τρία χρόνια για τη διαρθρωτική πολιτική και την κριτική που γινόταν σε ό,τι αφορά τη γεωργία και την αλληλεία ε, είχαν ε, ε καταλήξει ε, είχαν όμως βάλει στην πρώτη γραμμή του πυρός τη διαρθωτική πολιτική. Σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή πρέπει να αρχίσει μια συζήτηση που θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ίσως και στην Ολομέλεια πρέπει να γίνει. Αλλά ή δυνατόν όχι στις 11.30 το βράδυ στο Στρασβούργο, αλλά να ε, γίνει ε, την κατάλληλη ώρα. Κάνουμε κοινέ συζητήσει για θέματα λιγότερο σημαντικά σε πολύ καλές χρονικές ε, στιγμές, σε καλούς χρόνους για την πολιτική συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική που είναι τόσο σημαντική για όλη την Ευρώπη και τις περιφέρειες, χρειάζεται επίσης μια καλή συζήτηση. η Κωνσταντσή και μετά ο Λάμπερτ. Να απαντήσω σύντομα στον συνάδελφο προκειμένου περί του δημοσιονομικού πλαισίου έχεις δίκιο γιατί πραγματικά ε, έχουμε κολλήσει αλλά προκειμένου περί της διαπραγματευτικής εντολής και τα θέματα περιεχομένου ουσίας για την πολιτική συνοχής η εντολή της Προεδρίας που, τη βλέπουμε στην Κορεπέρ είναι πολύ μεγαλύτερη, πιο περιεκτική από ό,τι ε, ε, διαπραγματεύονται εκείνοι. Η Προεδρία δεν έχει υποβάλει έκθεση. Τα κράτη-μέλη δεν ξέρουν πόσο έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση και τις τελευταίες εβδομάδες αυτά που έγιναν δεν τα γνωρίζουν. Εμείς βέβαια ε, Προφανώς έχουμε ε, επαφές και με άλλα μέλη από το Συμβούλιο και ε, μας λένε ότι μπορείτε να κάνετε διαπραγματεύσεις και η Προεδρία έχει εντολή για διαπραγματεύσεις, απλώς ε, έχει διαφορετική στρατηγική η Προεδρία. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Κυπριακής και Ιρλανδικής Προεδρίας. Γιατί όλοι πιστεύαμε ότι με τους Κυπρίους δεν θα είχαμε προχωρήσει πολύ αλλά ο στρατηγικός σχεδιασμός ολοκληρώθηκε σε επίπεδο που δεν το πιστεύαμε ότι θα ήταν δυνατό να γίνει. Είχαμε κώδικα δεοντολογίας, είχαμε πάρα πολλά πράγματα ε, που προχωρήσαμε ενώ θεωρούσαμε ότι δεν θα τα τελειώναμε. Ενώ η Ιρλανδική Προεδρία τα σκέφτεται επί μήνες, διστάζει, καθυστερεί για να μας ε, ε, ασκήσει πίεση ε, για να ακολουθήσουμε στο τέλος την πρόταση της Προεδρίας και να μην προβάλλουμε τις δικές μας αξιώσεις. Αυτό είναι που μας έφερε στην τωρινή κατάσταση. Εμείς πάντως θα διαπραγματευτούμε όσο γίνεται περισσότερο και βεβαίως θα έχουμε υπόψη μας και τις συμβιβαστικέ λύσεις γιατί τον Οκτώβριο θα πρέπει να υπάρξει συνολική πρόταση για την πολιτική συνοχή στην Ολομέλεια και αμφιβάλλω αν ε, μέχρι τότε θα προλάβουμε να, να τα κλείσουμε όλα δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν τολμάω να κοιτάξω γιατί ψάχνω και δεν βλέπω κανέναν οπότε τι να κάνουμε να κλείσουμε τη συζήτηση. Α, Λάμπερτ, από ό,τι θυμάμαι ζητήσει το λόγο στα Ολλανδικά. Με τόσους με, με, τόσους και τόσους Να πω για αυτά που είπε η Κωνσταντσε τώρα έχουμε ε, τη διαδικασία ε, να συζητήσουμε, να κάνουμε και την ψηφοφορία στην Επιτροπή να επικοινωνήσουμε σχετικά με αυτά που έχουμε επιτύχει δεν ε, θα ανοίξουμε όλα τα θέματα που έχουμε επεξεργαστεί. Ε, ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει το τοπίο μέχρι τον Οκτώβριο και να μην έχουμε καμιά τρακοσαριά τροπολογίες, να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά θέματα και να κάνουμε συζήτηση για αυτά. Και στην Ολομέλεια θα γίνει επίσης αυτή η σημαντική συζήτηση, όπως είπες και εσύ. ούτως ώστε να δώσουμε ε, ε, μια πολιτική όθηση στην πολιτική ατζέντα μας στο Στρασβούργο. Λοιπόν, θα τα ξανασυζητήσουμε και αν έχετε κάποια θέματα, ελάτε, αναφέρετε τα στην Επιτροπή ή απευθεία σε εμάς. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Τότε, παρακαλώ, δώστε μου ένα πεντάλεπτο, ένα τρίλεπτο για να κάνω κάποιες ανακοινώσεις για την διαδικασία την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά πρώτα-πρώτα. Εγώ θα γίνουν τον, τον Ιούλιο αυτές, αυτή οι τερμινές διάλογοι, και είχαμε στείλει Γενικό Οργανισμό στο... κατά την Κυπριακή Προεδρία. Οπότε τώρα ίσως είναι πιο εύκολο, γιατί αυτό που τώρα και μόνο κανονισμό, αντίθετα με την αρχή, αλλά το θέμα είναι βέβαια ε, το ότι το πόσο ικανοποιημένοι θα είναι οι συνεισηγητές εξαρτάται από το μέγεθος καθαρά του γενικού κανονισμού που αποτελεί μια πρόκληση. Είναι τρομερό. Όλα είναι αλληλένδετα. Τεχνικές συνεδριάσεις έγιναν. Ήταν περίπλοκη διαδικασία και διαδρομή από την οποία τώρα βγαίνει η νικητής στο κοινοβούλιο. Δεν είναι θέμα το ότι κάνουμε υπήρξη δύναμη, αλλά περισσότερο ότι αυτό που μας καίει είναι η ποιότητα της πολιτικής την οποία διαμορφώνουμε. Έτσι όπως τα σιωπημένα τα βλέπω καμιά φορά και νομίζω ότι όλες οι πλευρές αυτό ήθελα. Πώς θα καταλήξουμε τελικά στην καλύτερη πολιτική. πάντως. Και τώρα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Αρχίσαμε τη βάση εντολή τη διαπραγματεύσει τον Ιούλιο και κατόπιν είχαμε ακόμα ε, μια συμπληρωματική διαδρομή ας πούμε ε, στην Επιτροπή Περιφερειακής ε, Πολιτικής κάθε φορά που έγινε μια καινούργια φάση σε αυτή τη διαδρομή κάθε φορά προσπαθούσαμε να λάβουμε ως βάση το που κατέληξαν οι κάθε φορά διαπραγματεύσεις. Οπότε έτσι υπήρξε αλληλοσυμπλήρωση των εντολών και των συζητήσεων. Έχετε λάβει τα εγγραφάκια για αυτή την συνάντηση θα πρέπει αυτό να το έχετε υπόψη, να το ξεχνάτε τώρα, όπως έλεγαν και οι δύο εισηγητές. Τέλη Μαΐου πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή, αυτή η διαδικασία, διότι έχουμε αυτή την έκθεση που θα έχει τότε ολοκληρωθεί και τότε θα στείλουμε το κείμενο για μετάφραση. Πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία στο Κοινοβούλιο. Στο μεταξύ δε θα ξεκινήσει η, να τρέχει προθεσμία για τις τροπολογίες. Τέλος Μαΐου θα έχει λήξει και μετά πάμε 12 με 20 Ιουνίου για την επόμενη, το επόμενο στάδιο. Οπότε και η γραμματεία πρόκειται να σας διαβιβάσει όλες τις ε, πληροφορίες, όλα τα τεχνικά τα οποία αφορούν την υποβολή των τροπολογιών. Ο Λάμπερ και η Κωνσταντζα μας εξήγησαν ότι θα πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα όσον αφορά τις τροπολογίες για τη διαδικασία αυτή, για την έκθεση αυτή. Βέβαια, όλοι θα μπείτε στον πειρασμό να δείτε τι γίνεται με τις τι γίνεται με τις τροπολογίες σας, οπότε εάν δεν καλυφθείτε, ίσως θέλετε τις ε, τροπολογίες να τις ε, αποσύρετε ή να εμείνετε αντίστοιχα Οπότε αυτό θα έχει μεγάλες επιπτώσεις. Γι' αυτό συνεργαστείτε με τους σκιώδεις ηγετές ο καθένας της πολιτικής του ομάδας, με τον συντονιστή σας, πριν την υποβολή των τροπολογιών για να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα των ε, επικαλύψεων και μετά να έχουμε απόρριψη τροπολογιών γιατί δεν θα υπάρχει αρκετή πλειοψηφία και ταυτόχρονα να απασχολείται την ε, ε, γραμματεία που εντατικά δουλεύει. 15 ώρες κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό. Και άμα φτάσουμε να έχουμε χιλιάδες τροπολογιών, ε, τότε υπάρχει υπερβολικός φόρτος εργασίας, δεν θα μπορούν να δουλέψουν έτσι τόσο ώστε να αποσπάσουμε το επιθυμητό πολιτικά αποτέλεσμα. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι το 100%. Ακόμα υπάρχουν πολλά προς διαπραγμάτευση. Αλλά να συγχυστούν οι διάλογοι. και ίσως και για τα νομιστικά κείμενα που έχουν κλείσει, ίσως ακόμα χρειάζεται να γίνουν για συγκεκριμένα σημεία κάποιες διαπραγματεύσεις και τον Ιούλιο θα γίνει η ψηφοφορία. Στόχος είναι μάλλον να πάμε για ψήφιση στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Σας είπα, για τη διαδικασία θα σας ενημερώσει η Γραμματεία. Και γενικότερα, ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να πεθυνθείτε στη Γραμματεία, στους και στους συντονιστές και έτσι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ούτως ώστε να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. από τι μου λένε η μετάφραση χωρίς να είναι σίγουρο θα έχει ολοκληρωθεί περί τις 14 Ιουνίου αλλά θυμηθείτε ότι οι τροπολογίες γίνονται επί του κειμένου της Κομισιόν οπότε έχουμε τις ε, διαπραγματεύσεις από την πρόταση της Κομισιόν και, την, και τις δικές τροπολογίες οπότε ελπίζω να θυμάστε να μην έχουμε τελικά παρά πολλές τροπολογίες. Κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Θα σας στείλει λοιπόν την τεχνική ενημέρωση της διαδικασία η, γραμματεία και μετά είπαμε ότι πάνε τα βοήθεια. Εγώ στην άλλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η τελευταία συνάντηση για τη διαλόγου έγινε 13 Μαΐου και έτσι μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί ολοκληρώθηκε η ιστορία αυτή, ο τριμερή διάλογος, ε, ε, εκκρεμώ αυτό που θα σας πω, απλώς, περιεχομένου τώρα. Δεν κάναμε τίποτα ε, ουσιαστικές αλλαγές, διότι βασικά θέλαμε να ευθυγραμμίσουμε το κείμενο του Ταμείου Συνοχής με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ένα σημαντικό πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, είναι αυτό το οποίο αφορά τους κοινού δείκτες, κάτι το οποίο είναι ε, θέμα το οποίο αφορά τον, τον οριζόντιο κανονισμό, τους άλλους κανονισμούς για το, για το Ταμείο Επικράτειας και τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα και είπαμε να πάμε για μια κατανάθεση κατ' σε πράξη. Αυτή να είναι η επιλογή μας και επίσης να έχουμε παράρτημα στον ε, κανονισμό σαν εναλλακτική λύση. Είπαμε επομένω να δοθεί, να, να ληφθεί η οριστική απάντηση στον τρίτο, διάλογο για τον κανονισμό για το περιφερειακό ταμείο ε, να σας πει ο Γιάννη επίσης αν θέλει πώς βλέπει τον, τον συμβασμό τον οποίο κλείσαμε. Επίσης ε, έχουμε τώρα αυτή την μακροοικονομική προϋπόθεση η αιρεσιμότητα ε, για το Ταμείο Συνοχής και συμφωνήσαμε με την Προεδρία ότι καλύτερα οποιαδήποτε τελική απόφαση για τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις να το αφήσουμε για τον τριμερή διάλογο όσον αφορά τις, ε, το, το, το, το ταμείο. Οπότε, οι αιτιολογικές παράγραφοι θα είναι ε, αντικείμενο έγγραφης διαδικασίας. Αν χρειαστεί να κάνουμε και συνεδριάσεις. Έτσι θα εξοικονομήσουμε κάποιο χρόνο και θα λάβουμε για τις αιτιολογικές παραγράφους την τελική απόφαση μόλις ε, όλα τα που ε, διεκπεριωθούν. Ακόμα και όπου έχουμε κάτι που αφορά το πολιτές δημοσιογραφικό πλαίσιο ή το CPR. Και με αυτόν τον τρόπο θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις όσον αφορά τον τεχνικό τριμερή διάλογο. Έχουμε την τροπολογία 15. Εκεί ζητούμε να έχουμε την ε, Euro Facility, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση, να τη συνδέσουμε με το κείμενο που αφορά το Κοινικό Ταμείο. Δεν άρεσε αυτό στο Συμβούλιο. Αν τελικά γίνει μεταφορά πόρων από το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Συνοχής στο Connecting Europe Facility, στη διευκόλυνση Connecting Europe, ε, αυτό δεν τους άρεσε να μπει στον τονισμό, αλλά τελικά συμφωνήσαμε και αποφασίσαμε όλα αυτά να μην ενταχθούν σε ένα άρθρο όσον αφορά το παιδί εφαρμογή, αλλά σε ενα καινουργιο καινούριο άρθρο 2α με μια υποσημείωση που να εξηγεί ότι αυτό το άρθρο θα πρέπει να ολοκληρωθεί όταν γίνει η τελική ρύθμιση ε, επί τη βάση του άρθρου 84 του κανονισμού για τις κοινέ διατάξεις. Οπότε εδώ συμφώνησε το Συμβουλίο όσον αφορά την τροπολογία 26 για την ε, ε, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος είπαμε να ευθυγραμμίσουμε τις διατάξεις μας με τις διατάξεις του ε, Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης να γίνουν επενδύσεις σε αυτό το κλάδο αλλά χωρίς αυτό να είναι η μόνη επιλογή. Όπως είπα και πριν, θέλουμε να υπάρχει η ευθυγράμμιση μεταξύ κανονισμού, ε, Ταμείου Συνοχής και Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης να γίνει συντονισμός των ε, διατάξεων, υπάρχει αντιστοίχηση και έτσι αυτό θα αποτελέσει απλούστευση για καλύτερη πρακτική και θα γίνει πιο εύχριστο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξήλθαμε όλα τα άρθρα εκεί που χρειαζόταν κάποια ευθυγράμμιση, ακριβώ όπως θεωρώ ότι έγινε στον και στον κανονισμό για το Περιφερειακό Ταμείο. Και σας τονίζω ότι αυτό είναι το κλειδί για μια πραγματική απλούστευση. Οπότε έτσι αλλάξαμε αργούς μεγάλες αλλαγές τι, τα, τα, μέτρα για, τα, για τις θεομηνίες οπότε και, και τώρα για το δυτικό τμήμα είπαμε ότι ήταν ε, δύσκολο να τηρήσουμε το περιβαλλοντικό κεκτημένο αλλά πάλι είπαμε ότι θα πρέπει να ισχύσουν κάποια στάνταρ, κάποια πρότυπα όταν ε, τα κράτη-μέλη και επισημάνουν τις ανάγκες τους. Τώρα, όσον αφορά την ανάγκληση του κανονισμού, είπαμε και πάλι για λόγους συνέπειας, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου ληφθεί απόφαση στα πλαίσια του κανονισμού των κοινών διατάξεων και θα ευεργαμιστούμε τότε με αυτόν. Όλα αυτά διεκπεριώθηκαν υπό την Προεδρία της Κανούτα. Οπότε θέλω να πω ότι η κυρία Χιούμνερ, ε, ευχαριστούμε πολύ, λέει στα πολωνικά. Συγγνώμη, συγγνώμη, τα κουτσά στραβά τα λέω στα πολωνικά. Τι να σας πω. Είδατε ξαφνικά διαμαγείας βελτίωσε στα πολωνικά μου. Θαυμάζω τον εαυτό μου. Να ναι, το είπα και για πολιτική ορθότητα, αλλά όντω η πρόεδρο βοήθησε πάρα πολύ. Και ο Νίκολα Μάρτιν και ο Πίτερ επίση βοήθησαν πάρα πολύ. Είχαμε επίσης διαρκή βοήθεια, υποστήριξη και ενώ στην αρχή βλέπαμε να μην υπάρχει περιθώριο λιμών, τελικά βρέθηκε ο συμβασμός. Τελευταίο αλλά σημαντικό, συγχαρητήρια και στους διαπραγματευτές και στην Ερμήνια και στη Ραμόνα, την Ρουμάνα συνάδελφο, και στον ε, Όλτριτς και στην Κορνιλία και στον Νίκολας. και στον Ιωσήφ δηλαδή διότι διακριτικά, αλλά πάρα πολύ μας στήριξε σε δύσκολες στιγμές. Σας ξαναευχαριστώ όλους. Τα καταφέραμε και τα καταφέραμε με έναν τρόπο που θεωρώ ότι θα ωφελήσει πάρα πολύ τις περιφέρειές μας, τις κοινότητές μας. Ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό σαν ε, πολιτικό έργο. Ε, γιατί ήταν ε, ε, πάρα πολύ αγαστή συνεργασία παρά το ότι προερχόντουσαν από διαφορετικές πολιτικές πτέρυγε οι συνεργαζόμενοι. Ήταν ε, μια διαδρομή που επίσης παρακολούθησαν και τα εθνικά μας κοινοβούλια και έτσι αποδείχθηκε ότι για την πολιτική συνοχή τουλάχιστον εδώ υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν καλά και επιδέξια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πρόεδρος και τώρα αν θέλετε να συζητήσουμε. Αλλά ίσως έτσι κατάλαβε ο Επιτροπή ότι τόσο πιο εύκολα διεκπληρώνουμε τα πράγματα, όσο πιο μικρό είναι το κείμενό σας. Δεν θέλει κανείς το λόγο. Α, θέλει και ο Σόλμπριτς. Και ο ναι. ε, όχι, δεν μπορεί να γλύσει έτσι η συζήτηση, Βίκτορα. Όχι απλώ θέλω να δούμε τι γίνεται με αυτά τα δέκα δις τελικά. Έχουμε συμφωνήσει για την ημερομηνία. Τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα. Ο συμβασμός ε, όπως έκλεισε αφορά το, σαν κατελήτη ημερομηνία Δεκέμβριο του 2016 Ιανουάριο του 2017 για να δούμε λοιπόν αν περισσεύουν ακόμα χρήματα, τότε πρόκειται να μεταφερθούν στην κεντρική διαχείριση ε, της, ε, της διευκόλυνσης. Connecting Europe. Και έχουμε τώρα και τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές πλαίσιο, οπότε και τα χρήματα πρόκειται να διατεθούν από εκεί, στο Connecting Europe. Αλλά δεν είμαστε πεπισμένοι ότι τελικά θα δοθούν τα χρήματα αυτά τα οποία πρότεινε τον Φεβρουάριο το Συμβούλιο. Γιατί αν δεν υπάρξουν τα χρήματα που πρέπει, αυτά που είχαν προβλεφθεί, τότε δεν έχει νόημα η διευκόλυνση. Εδώ και προτείνω αυτό το συμβασμό και είπαμε να μην αναφερθούν συγκεκριμένα νούμερα. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με βρυκοδότηση, Χωρίς βρυκοδότηση και μόνο με τα 10 δις του, γραφείου, του Ταμείου Συνοχής ε, δεν έχει νόημα. Δεν θα έχει επιπτώσεις σε σχέση με την ε, διασυνοριακή διάσταση ε, αυτών των προγραμμάτων για τη συμφωνία. Ε, πρόεδρος. Προς το παρόν δεν υπάρχει δεκάρα, ούτε τα δέκα δις. για δεν θέλετε να συζητήσουμε κάτι άλλο, σας πενθυμίζω ότι η γραμματεία ε, ελπίζουμε Μία Μαΐου, 1η Ιουνίου να έχει τα, τις μεταφράσεις και όπως είπαμε και πριν 12 με 20 Ιουνίου θα πρέπει να προβληθούν τροπολογίες δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει ή όχι αύριο πάντως θα έχουμε τον Επίτροπο Αλμούνια και έχουμε ακόμα διευθυντικές γραμμές όσον αφορά αυτή την διαβούλευση μεταξύ των υπηρεσιών. Οπότε έχουμε να συζητήσουμε ένα σωρό ζητήματα με τον Επίτροπο. Ενέργεια, υποδομές, ε, ηλεκτρική ενέργεια και την παραγωγή της. Όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα οπότε ελάτε αύριο με πολλές ερωτήσεις προς τον Επίτροπο Αλμούνια για να δούμε πώς αυτές οι μεγάλες υποδομές θα προχωρήσουν και πώς θα καλυφθούν από τις κατευθυντήριες της περιφερειακής βοήθειας. Τώρα, ο Γιάννη έχει το λόγο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι διαπραγματευόμαστε ένα πολύ μεγάλο ε, κείμενο το οποίο συμβαδίζει βεβαίως από, με τη συνθήκη από όσο γνωρίζω. Όσον αφορά το, τους τριμερείς διαλόγους για το ΕΤΠΑ, είχαμε 13 στον αριθμό και υπάρχουν γενικά σχόλια που πρέπει να γίνουν. Θα ήθελα να τονίσω το ρόλο της δύναμης, της ομάδας διαπραγμάτευσης που έχει διτό ρόλο. Διαπραγματευόμαστε καταρχήν μεταξύ μας και εδώ είναι το πρόβλημα διότι έχουμε μία εντολή και δεν ξέρουμε πόσο μπορούμε να προεκταθούμε από το είναι εντολή και γίνονται σκληρές συζητήσεις ε, μέσα στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει και στη συνέχεια έχουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με την παρουσία της Κομισιόν μετά από τις εσωτερικές μας ε, διαπραγματεύσεις. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω διότι δεν θέλουμε να ε, επανέλθουμε με τις ε, τροπολογίες όπως ήδη προελέχθη. Ένα άλλο θέμα που μας εκπλήσει κάπως και μένα ως εισηγητή είναι η ασυνέπεια των νομικών υπηρεσιών των τριών θεσμικών οργάνων. Αυτό πρέπει να αναφερθεί και να αναφέρεται σε όλες τις εκθέσεις. Έχουμε μία ενωμένη Ευρώπη και τρία βασικά θεσμικά όνα και υπάρχουν και οι διαθεσμικές συμφωνίες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διάφοροι ε, νομομαθείς που μπορούν να ερμηνεύσουν διαφορετικά τις συνθήκες. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε νομικές υπηρεσίες που ε, πολεμούν οι μεν τις δε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς είμαστε πολιτικοί και θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές μήνυμα από τη νομική υπηρεσία. Όχι να έχουμε αυτό το παιχνίδι μεταξύ νομικών υπηρεσιών όπου μας διαγωνίζουν οι μεν και οι δε γιατί φτάσαμε και στο σημείο ένας δικηγόρος να μας πει θα σας ε, ε, θα κάνω, θα κάνω μήνυση. Θα σας κάνω μήνυση. Γιατί οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι της Κομισιόν λένε ότι θα κάνουν προσφυγή στο δικαστήριο. Ποιος θα το κάνει, θα το κάνει ο Μπαρός, θα το κάνει ο Φανορόμποη. Αυτό είναι απαράδεκτο να γίνεται λόγος για προσφυγές. Οι νομικές υπηρεσίες πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Για να υπάρχει μία και μοναδική ερμηνεία της συνθήκης διαφορετικά, είναι πολύ επικίνδυνο. Σημαίνει ότι οι πολιτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νομικές υπηρεσίες για να παίξουν δικό τους παιχνίδι ο καθένας από μας μπορεί να προβάλλει και τη γνώμη μιας νομικής υπηρεσίας από τη χώρα μας, για να έχουμε ακόμα περισσότερα επιχειρήματα υπέρ ημών. Αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο, δεν μπορούμε να το δεκτούμε. Ως προς το περιεχόμενο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που διέπουν το ΕΤΠΑ, Φτάσαμε σε μια συμφωνία μετά από δύσκολες συζητήσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και ως προς το θέμα της επιλεξιμότητας έγινε λόγος για μεγάλες επιχειρήσεις για ΜΜΕ αλλά και ε, για τις υποδομές, ε, για τις βασικές υπηρεσίες στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές. Φτάσαμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο και το επιβεβαίωσε και η Κομισιόν. Ήταν πολύ δύσκολη η συζήτηση και για τις προτεραιότητες, τις επενδυτικές ε, προτεραιότητες, τους θεματικούς στόχους και έχει επέλθει συμφωνία και υπάρχει και το νέο στοιχείο της αστικής διάστασης που πρότεινε η Επιτροπή, δηλαδή η παρέμβαση στα μεγάλα αστικά κέντρα και οι ενωμένε ε, δράσεις ε, για τα μεγάλα αστικά κέντρα με βάση και τις, ε, την, τις νέες τεχνολογίες και την, και την πληροφόρηση για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο αλλά έχει συμφωνηθεί. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που παραμένουν ανοιχτά. Η θεματική συγκέντρωση. Αυτή η θεματική συγκέντρωση, σε αυτή την θεματική συγκέντρωση φτάσαμε στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες, αυτές που είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και την ειδική μεταχείριση για την Ιρλανδία. Έχουν ε, συμφωνηθεί όλες οι διαστάσεις του θέματος. Υπάρχει και ένας μηχανισμός αντιστάθμισης που προσδίδει στα κράτη-μέλη τις δυνατότητες για να αλλάξουν τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα. Πρόκειται για ένα ευέλικτο μέσο, συμφωνούμε για τη θεματική συγκέντρωση και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν ό,τι επιθυμούν. Πρόκειται για ένα μηχανισμό αντιστάθμισης. Συμφωνήσαμε όμως γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά για μας. Ε, τα θέματα που σχετίζονται και με το ΕΚΤ και το θέμα αυτό σχετίζεται και με τη θέση του Συμβουλίου. Διότι μας είπε το Συμβούλιο ότι δεν θα φτάσουμε στη θεματική συγκέντρωση αν δεν συμφωνήσει και το ΕΚΤ. Ελπίζουμε λοιπόν να δοθεί τελική μορφή σύντομα, γιατί αν αλλάξει κάτι στο ΕΚΤ, στοιχεία δηλαδή που μπορεί να πειράσουν το όλο σύστημα, θα πρέπει να ξανανοίξει ολόκληρο το πακέτο της, των, της θεματικής αυτής, της θεματικής συγκέντρωσης. Νομίζω ότι η Επιτροπή παγιδεύτηκε ένα από τα βασικά μας ερωτήματα προς την Επιτροπή, που ίσως θα θυμόσαστε, είναι αν έχουμε 7 θεματικούς στόχους, ποιοι προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ποιοι, ποιες θεματικές ενότητες από τις 11 προέρχονται από το ΕΚΤ. 8, 9 και 10 είναι για το ΕΚΤ και για το ΕΤΠΑ οι υπόλοιπες, οι 11. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επικάλυψη σε τρεις θεματικούς στόχους και εδώ επικεντρώνεται η συζήτηση για την επικάλυψη για, τους, ε, για τις θεματικές ενότητες 8, 9 και 10, όπου υπάρχει επικάλυψη των δύο ταμείων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα, θα έπρεπε να δούμε τι θα έπρεπε να έχει ανατεθεί στο ΕΤΠΑ και τι στο ΕΚΤ. Αλλά τώρα είναι πολύ αργά και το πρόβλημα είναι η επικάλυψη. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να συγκεντρωθούμε στις θεματικές ενότητες ή στα επιμέρους θέματα. Ε, τελειώσαμε τις συζητήσεις για τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια, τις τέσσερις ενότητες, τις τέσσερις πρώτες. του θεματικού αυτού στόχους, τους πρώτους τέσσερις δηλαδή. Κάτι το οποίο μας εξέπληξε, αλλά ίσως ε, δεν εκπλήσει αυτούς που γνωρίζουν, ε, δεν ε, προβληματίζει αυτούς που ξέρουν πολύ καλά τις συνθήκες, δηλαδή η κατεξουσιοδότηση πράξη σε σχέση με τις εκτελεστικές πράξεις. Το ζήτημα είναι πώς θα εφαρμοστεί το όλο πλαίσιο με κατεξουσιοδότηση πράξης ή με εκτελεστικές πράξεις. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή πάνε στα πιο καυτά σημεία, δηλαδή οι καινοτόμες δράσεις που είναι σαφείς για μας. Είναι δράσεις που αφορούν την Κομισιόν. Δεν έχουν να κάνουν με τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να ισχύουν η κατεξιοδότηση πράξης αλλά το Συμβούλιο δίνει μεγάλη μάχη για να θεωρηθούν εκτελεστικές πράξεις. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται αυτό. Επίσης για τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές γίνεται μεγάλη, δίνεται μεγάλη μάχη. Εμείς έχουμε εισαγάγει την τροπολογία για τη ε, διαδικασία απλούστευσης, απλοποίησης για τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Και εμείς το υποβάλαμε σαν απλή τροπολογία αλλά έγινε μεγάλη συζήτηση για την λεγόμενη operating aid. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό έγινε λόγος και για προσφυγή. Από πλευράς χρημάτων είναι αμεληταίο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν οι νομικές υπηρεσίες μεταξύ τους. Σας το λέω αυτό, διότι αυτό είναι ένα ε, μικρό σημείο αλλά η συζήτηση είναι ύψη της σημασίας. Δηλαδή, αν ανοίξουμε αυτή την πόρτα, μπορεί να ανοίξει και αλλού και για τη κατεξουσιοδότηση πράξη. Ω προς τους δείκτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφους για τη θετική τους προσέγγιση, γιατί υπήρχαν δύο δυνατότητες εξ αρχής είτε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους ε, δείκτες από πολιτικής ε, άποψης, γιατί ξέρουμε πώς να τους καταρτήσουμε, και άλλοι είπαν ας μην τους αγγίξουμε όπως ο εισηγητής γιατί οι εμπειρογνώμονες θα το χειριστούν υπάρχουν ε, τεχνικά στοιχεία θέματα επαλήθευσης και αξιολόγησης δεν το αγγίξαμε και πάλι ήταν το θέμα κατά πόσο πρόκειται για μια κατεξουσιοδότηση, πράξη, εκτελεστική ή εντάσσεται στα παραρτήματα. Εμείς είπαμε ότι εντάσσεται στα παραρτήματα που δεν θα αλλάξουν τώρα, δεν θα τροποποιηθούν τώρα, θα βασιστούν στην πρόταση της ε, Επιτροπής όπως την είχε προετοιμάσει την πρόταση Επιτροπή εδώ και δύο χρόνια με τους εμπειρογνώμονες, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων. Δεν θα υπάρξει πλήρης αλλαγή, αλλά θέλουμε να σταθεροποιήσουμε κάπως την κατάσταση έτσι ώστε οι τελικοί δικαιούχοι να γνωρίζουν ότι ε, ε, ο δείκτης αυτός είναι διαχρονικός. Υπάρχει από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μικροαλλαγές με κατεξουδότηση πράξης μόνο. Συνοψίζοντας, παρά τις δυσχερείς διαπραγματεύσεις και στην ομάδα, γιατί και εδώ ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις και αυτό σήμαινε ότι οι σκιώδεις πρέπει να φτάσουν σε συμβιβασμό. Και αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Και αν έχουμε τη συμφωνία και του ΕΚΤ, τότε θα ψηφιστεί το θέμα τον Ιούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον Γιάννο Όλμπριχτ για την πορεία που έδωσε στο θέμα. Καλό είναι που συζητήσαμε στη διαπραγματευτική ομάδα και είχαμε μια σχετική ε, ομοφωνία, ομόφωνη γνώμη στον τριμερή διάλογο και κλεισμένο των θυρών. Και γι' αυτό καταφέραμε αυτά που καταφέραμε. Σε κάποιους τομείς, στους 11 θεματικούς στόχους, θέλαμε κάτι παραπάνω. Και αυτή ήταν και η βάση με την οποία πήγαμε στις διαπραγματεύσεις. Α, δεν τα καταφέραμε, αλλά κάναμε τις λιγότερες υποχωρήσεις. Σε πολλά θέλαμε κάτι παραπάνω, αλλά με το αποτέλεσμα που πετύχαμε νομίζω την περασμένη Δευτέρα, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να δηλώσουμε ικανοποιημένοι. Θυμάστε την υπόθεση με το αέριο που συζητήσαμε με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση στην αιτιολογική σκέψη δεν αναφέρεται ακόμα το αποτέλεσμα που πετύχαμε τη Δευτέρα Τώρα ε, θα πρέπει το, η λέξη αέριο να αντικατασταθεί από τη λέξη ενέργεια και αυτό θα γίνει δεκτό. Ή θυμίζω τη συζήτηση για τα λιμάνια που την πήγαμε μέχρι το τέλος, αν θα κατασκευαστούν ή όχι. Γενικά Πάντα έτσι γίνεται στις διαπραγματεύσεις. Σε ορισμένα πράγματα είπαμε όχι, αλλά εμείς, ε, η ομάδα του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους πολίτες, έκανε το καλύτερο δυνατόν. Και καταφέραμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Για την Προεδρία ακούσαμε πολλά. Οι διαπραγματεύσεις πάντως ήταν σκληρές. Στον πρώτο τελευταίο ε, τριμερή διάλογο ξεκαθαρίσανε λίγο τα πράγματα και είπαμε που μπορούμε και που δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ προβληματίστηκα από αυτό και Νομίζω ότι καλά κάναμε γιατί εμείς το οφείλουμε στους πολίτες να δηλώνουμε ότι είμαστε ισότιμος εταίρος. Αυτά λοιπόν που μπορούσαμε να καταφέρουμε, τα καταφέραμε. Ευχαριστώ. Και εγώ επιβεβαιώνω ότι οι Σκιώδη ήταν πολύ δραστήριοι σε αυτό το τριμερή διάλογο. ναι, ήταν πολύ δραστήρι και θετική. <laughs> Άλλα σχόλια υπάρχουν. Κύριο Σόλτριξ, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ αισθάνομαι ικανοποιημένο για το συμβασμό. Τέλεια. Όμως, νομίζω ότι υποκρύπτεται κάποιος κίνδυνος στις λεπτομέρειες άρα θα πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ προσεκτικά όσον αφορά την κατεξιοδότηση πράξη και τις λεπτομέρειες Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι, με προσοχή και επίσης σε σχέση με την υποστήριξη των μεγάλων εταιριών. Έχουμε τις προϋποθέσεις ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνει συνεργασία με ΜΜΕ, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιο είναι το περιεχόμενο, τι σημαίνει αυτό. Να κινηθούμε με μεγάλη προσοχή. Και τελικά αισθάνω μεγάλη ικανοποίηση γιατί όλες οι προϋποθέσεις που έχω τάξει έγιναν δεκτές και άρα δεν μπορώ παρά να σας συγχαρώ όλους. Ευχαριστούμε λοιπόν Πρόεδρος. Άλλες ε, παρατηρήσεις. Οπότε και εγώ θα πρέπει να επαναλάβω την ίδια πρόταση. Η δε ε, γραμματεία θα σας στείλει αυτή την ε, επιστολή και το 12 με 20 Ιουνίου θα υποβληθούν αυτέ τι τροπολογίε και πρέπει να σα πω ότι από τον κύριο Λαμασούρα έλαβα σήμερα τι πληροφορίε ότι αύριο στις 9 όπου έχουμε την συνεδρίασή μα αλλά και τον κύριο Αλμούνια στις 9 λοιπόν θα έχουμε τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι στην Επιτροπή των Προπολογισμών όπου και θα γίνει ενημέρωση για τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια ε, σαν ανάλυση του προπολογισμού. Οπότε, δεν μπορούμε να πάμε. Ούτε εσείς μπορεί να πάτε, αλλά μπορείτε να στείλετε κάποιον συνεργάτη. Επίσης έχουμε και την ε, γραμματεία μας που θα παρακολουθήσει και θα λάβουμε υπόψη ότι ε, ενδιαφέρον προκύψει. Πάμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Επόμενη έκθεση είναι η έκθεση της Ρίκα Ακάρινεν. Άλλαξε το όνομά της. Πακαρινέν Μάνερ τώρα. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία είναι σε αδιαμητρότητος. Ευχαριστώ όλους που συμμετέχουν στην τριμερή διάλογο για, ε, τη συνεργασία τους για, και για την υποστήριξή τους κατά διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά δε τον εν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτικής συνοχής η ευρωπαϊκή συνεργασία έχει ε, αυτό το καινούργιο πλαίσιο ε, νέα πολιτική και θα θυμάστε ότι η βασική μας ε, θέση στην εντολή ήταν ότι απαιτείται το να υπάρξει εδαφική συνεργασία στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Και έχουμε την πολιτική απόφαση του Φεβρουαρίου για το 7%. Και σε συμφωνία με τη Ρίκα, τότε, όταν ολοκληρώθηκε ο δεμερής διάλογος, αφήθηκε να επιστολή στον κύριο Σούλτ, τον πρόεδρο Σούλτ. Και του είπα ότι αν τυχόν η συζήτηση για τον προπολογισμό, να υπάρχει αυτή η εντολή από την Επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξη για να αυξηθεί η πρικοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Θα έπρεπε να πω ότι δεν πιστεύω ότι θα ξανανοίξει αυτό το θέμα. Αλλά είπαμε ότι έτσι θα μπορούσαμε να μετακινήσουμε κάποιους πόρους από την πολιτική πυρήνα προς την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Πέραν και των συμφερόντων της ε, κάθε χώρας. Να δούμε αν θα τα βρούμε το Συμβούλιο. Οπότε και έτσι θα προκύψουν οι πόροι που είναι βασικοί για αυτή την πολιτική. Έχουμε επίσης και τον κανονισμό που καλύπτει το θέμα της συμμετοχής των τρίτων σε αυτή την πολιτική. Οπότε πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους συνεργάτες μας γιατί ε, πάρα πολύ θετικός για το κοινοβούλιο αυτός ο συμβασμός. Επίσης έγιναν μακρές συζητήσεις σε μια σειρά τριμερών διαλόγων για διάφορα σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ETC, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Νίκολας, διόρθωση με κανενα λάθος και είπαμε ότι αυτό θα γίνει με χρηματοδότηση αναπρόγραμμα ή θα μπορούσε να γίνει με χρηματοδότηση ανά κράτος μέλος. Τελικά η πρώτη λύση επελέγει. Βέβαια τα κρατη με και έχουν το, το, το, τον προϋπολογισμό προτιμούν να έχουν τον έλεγχο. Οπότε γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι για την ε, δευτική συνεργασία θα έχουμε την χρηματοδότηση ανά κράτος μέλος. Και έτσι βέβαια είχαμε μια μικρή απογοήτευση στην διαπαντευτική ομάδα. Επίσης, Είπαμε να υπάρχει για την θεματική συγκέντρωση κάποια ευελιξία, όπως και στη συζήτηση του οργανισμού του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και τελικά το 80% για τους θεματικούς στόχους και ευελιξία για το υπόλοιπο 20%. Επίσης, να υπάρχει ευελιξία μεταξύ των δύο πτυχών της εδαφικής συνεργασίας. σε σχέση με το 15%. Άρα, είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα που αποσπάσαμε αυτό το συμβασμό. Και για την τεχνική αρρωγή. Η τεχνική αρρωγή είχε ζητηθεί περισσότερη ευελιξία. Όποτε η υλοποίηση απεδεικνύεται δύσκολη. Και εκεί επομένως είναι ικανοποιητικό το ότι κλείσαμε το συμβασμό. Για, τα, για τις τώρα αναλύουμε την πρόταση θα προχωρήσουμε με την ε, ε, έγγραφη διαδικασία όπως συνήθως με τους κανονισμούς. Ξεολόγηση του εισηγητή είναι ότι ως επιτοπλίστων έγινε ό,τι προέβλεπε η εντολή. όπου δεν τηρήθηκε η εντολή αυτό έγινε για καλό. Και έτσι λοιπόν διαχειριστήκαμε αυτά τα δύο ζητήματα, δηλαδή το επίπεδο της ε, στήριξης και την χρηματοδότηση ανά κράτος μέλος ή ανά πρόγραμμα. Θα ενημερωθείτε, θα σας διαβιβάσουμε την έκθεση Είπαμε τροπολογίες μεταξύ 12 και 20 Ιουνίου. Και μας έχει απομείνει τώρα μόνο η εκθέση του Γιώκημ. Μου είπαν ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελευταία περίοδο αυτός ο κανονισμός για τη ομίλους ήταν ο δυσκολότερος και τον διαπραγματεύτηκαν τελευταίο. Βεβαίως, μη πρωτού τέλους μακάριζε λέει κανείς. Είμαστε πάντως τώρα στην παραμονή. Την προπαραμονή έγινε ο τρίτος τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο και το κείμενο και τα άρθρα του κανονισμού έχουν συμφωνηθεί όσα έχουν νομική σημασία. Αυτό που λείπει είναι οι αιτιολογικές σκέψεις που θα μας έρθουν απόψε το βράδυ. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω επειδή καταφέραμε με τρεις διαπραγματεύσεις να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ την Πρόεδρο Πρωτίστως η οποία γνωρίζει πολλά και τάχθηκε υπέρ του Ευρωπαϊκού Ομίλου, τη Γραμματεία, τον κύριο Κάλιτα που είναι ο σύμβουλός μας και τον κύριο Ράιχελ τον, βοηθό μου που όλοι συνεργάστηκαν εξαιρετικά μεταξύ τους ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Κομισιόν, στους κυρίους Μάρτιν και Πέτερς που συνεχώς και με συνέπεια μας υποστήριξαν και όταν υπήρχαν δυσκολίες ε, βοηθούσαν και με συγκεκριμένη διατύπωση και απέδειξαν ότι στηρίζουν πολύ αυτό το νομικό μέσον. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ιρλανδική Προεδρία σε αυτό το σημείο, διότι ήδη πριν από την Ιρλανδική Προεδρία είχαμε κάνει άτυπες συνομιλίες με τους εκπροσώπους της Ιρλανδίας και μεταξύ των επισήμων τριμερών διαλόγων όταν υπήρχαν δυσκολίες στις επίσημες συνομιλίες ατύπως μπορούσαμε να συναντώμεθα. Είπα πριν ε, για τα κράτη-μέλη, ε, γνωρίζουμε, γνωρίζαμε τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, πολλές φορές διήσταντο οι απόψεις και οι δυσκολίες των Ιρλανδών είναι κατανοητές. Ήταν δύσκολο να τα συγκεράσουν, να συγκεράσουν όλες τις διαφορετικές απόψεις. Εν τω μεταξύ μας πέρασε η σκέψη ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν θα καταφέρναμε να υλοποιήσουμε το στόχο να ε, τελειώσουμε πριν από το καλοκαίρι. Τώρα φαίνεται ότι τα καταφέραμε. Περί τίνος πρόκειται, εμείς ε, κινηθήκαμε στα πλαίσια της εντολής που μας είχε δώσει η Επιτροπή και πρέπει να πω ότι είμαστε σε συνεχείς επαφές με τους πραγματικούς χρήστες ε, αυτού του μέσου, δηλαδή την Επιτροπή των Περιφερειών. Συνεχώς δηλαδή ε, κάναμε ε, διαβουλεύσεις σχετικά με κάποιες συμβιβαστικές διατυπώσεις και αν αυτές θα ήταν δυνατόν να γίνουν αποδεκτές από τους ε, χρήστες αυτών των ομίλων. Τώρα, ποια ήταν τα ιδιαίτερα σημεία που έχριζαν διαπραγματεύσεων εμείς με την επεξεργασία αυτού του κανονισμού θέλαμε να απλοποιήσουμε τον κανονισμό, να επιτύχουμε νομική ασφάλεια, μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του κανονισμού για τους ομίλους. Τα πιο σημαντικά ήταν ε, η ε, σιωπηρή έγκριση, τα approval, ε, αν δηλαδή η αρχή ε, έγκρισης ε, δεν αντικατοπτρίζεται, δεν δεν τον ε, όμιλο ή σιωπηρή συμφωνία για την δημιουργία νέων ομίλων μετά την λήξη της εξάμηνης περίοδου τότε θεωρείται ε, σιωπηρά δεδομένη. Υπάρχει μια εξαίρεση για το κράτος μέλος στον οποίο θα έχει την έδρα του Ευρωπαϊκού Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας. Θα πρέπει να συνεργάζονται περισσότερα κράτη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, το κράτος μέλος όπου θα είναι η έδρα πρέπει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες. Γι' αυτόν θα ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να τηρούν την εξάμεινη προθεσμία για το ε, ε, αλλά για το κράτος ε, που θα έχει την έδρα του ο Ευρωπαϊκός Όμιλος εκεί υπάρχει μια εξαίρεση. Νομίζω ότι οι επίπονες και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον Όμιλο απλουστεύονται ε, οι αυθαίρετες καθυστερήσεις ε, δεν θα είναι δυνατές. Η νέα ρύθμιση υποστηρίζεται και από μια κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Κομισιόν ε, και αυτή η δήλωση λέει ότι τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να τηρήσουν μια διαφανή διαδικασία και με βάση αυτά ε, θα προσανατολίζονται και θα πορεύονται και όσοι θέλουν τέτοιους ομίλους. Τώρα, ένα άλλο θέμα ήταν η εργασιακή νομοθεσία που θα ίσχυε για το προσωπικό. Μέχρι τώρα ήταν επίμαχο το θέμα αυτό. Και εδώ, στα πλαίσια των διαβουλεύσεων, ε, ε, παρουσιάστηκαν πολλές δυσκολίες πρακτικές. Υπήρχε δυνατότητα επιλογής δικαίου ε, αλλά αυτό συχνά ε, δεν ήταν γνωστό. Εμείς με την Κομισιό και το Συμβούλιο είπαμε να κάνουμε μια νέα δήλωση για να ε, αναφέρουμε το άρθρο που θα ίσχυε. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος θα μπορεί να εφαρμόζει το εργατικό δίκαιο που επιθυμεί για το προσωπικό του, θα μπορεί να επιλέγει και έτσι μια υφιστάμενη δυσκολία γιατί η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ομίλου έχει πλέον αρθεί. Επόμενο μεγάλο σημείο ήταν η συμμετοχή δημοσίων ε, δημοσίων φορέων ε, γενικού συμφέροντος, public services, δημοσίων υπηρεσιών. Τις τροπολογίες μας ε, τις στηρίξαμε στον κανονισμό που αναφέρεται σε αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες η αναφορά έλειπε στην αρχική πρόταση της Κομισιόν και εμείς ε, το είδαμε αυτό, είμαστε υπεύθυνοι για τις περιφέρειες, οπότε έγινε προσθήκη στον κανονισμό. Έτσι στο μέλλον και οι τομείς υγεία, παιδεία, εκπαίδευση, κατάρτιση και κοινωνικά θέματα συμπεριλαμβάνονται στη δυνατότητα ίδρυσης ομίλων, Διασυνοριακά ε, ε, νοσοκομεία και βρέφονιπιακοί σταθμή δεν έχουν πια προβλήματα. Ε, ανάλογα με την εντολή μας διαπραγματευτήκαμε ότι στο μέλλον μόνο η ε, σύγκληση πρέπει να εγκρίνεται χωριστά. Αυτό ε, σημαίνει ότι το καταστατικό ε, δεν χρειάζεται ειδικό κανονισμό γιατί αφορά την εσωτερική λειτουργία του κάποιου ομίλου και δεν αφορά την ποιότητά του εις ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών. Άρα λοιπόν ε, είπαμε ότι μόνο η συμφωνία για την ίδρυση του ομίλου χρειάζεται έγκριση και μετά κοινοποιείται ο εσωτερικός κανονισμός που δεν χρειάζεται να εγκριθεί και αυτός. Ένα άλλο σημαντικό σημείο ήταν, και αυτό είναι καινούριο στοιχείο, προκειμένου περί ιδρύσεων ομίλων, είναι η συμμετοχή τρίτων χωρών. Εδώ ε, βρήκαμε έναν ε, ευρύ και ε, σαφή ορισμό ε, σχετικά με την επαφική συνεργασία με τρίτες χώρες. Επίσης οι εξόχως μακρισμένες περιοχές, τα υπερπόντια εδάφη ε, πρέπει να εξεταστούν ε, γιατί η ίδρυση ομίλων δεν ε, έχει να κάνει με μεγάλες αποστάσεις, είτε είναι η Μαδέρα είτε η Καταγανάρια νησιά, μπορούν και εκείνοι να ιδρύουν τέτοιους ομίλους. Η θάλασσα δηλαδή δεν ισχύει ως ε, ε, σύνορο. το αναφέραμε και αυτό στο κανονισμό, ότι υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ίδρυσης τέτοιων ομίλων και αυτό πιστεύω ότι είναι άλλο ένα βήμα μπροστά. Ελπίζω ότι το πακέτο που ετοιμάσαμε θα διατηρηθεί, δεν θα αλλάξει. Περιμένουμε και τις αιτιολογικές σκέψεις που τις έχουμε συζητήσει και δεν χρειάζεται να κάνουμε έξτρα τριμερή διάλογο για αυτές. Ε, μπορούμε δια της γραπτής διαδικασίας να τελειώσουμε το κομμάτι αυτό, ούτω ώστε να τεθεί σε για ψηφοφορία όλο το πακέτο. Και ελπίζω ότι θα, έχω θα έχουμε την θετική σας ψήφο. Και πάλι ε, να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν. Μαρή Τερέζα. Ας με συγχωρήσει ο Γιώκεμ, αλλά συστηματικά παίρνω τον λόγο ως σκιώδες για την δευτική συνεργασία. Οπότε να σας πω δύο λόγια. Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις. Βέβαια θα πρέπει να δούμε οριστικά να κλείσουν και οι λόγια παράγραφοι όσον αφορά τώρα τον προπολογισμό. Μην θεωρήσουμε ότι έχει χαθεί η μάχη τη ευθύ εξ αρχής στην έκθεσή μου εδώ και δύο χρόνια ή ε, σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε, ζητάμε την αύξηση και θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη μας από αυτού γιατί εάν υποχωρήσουμε πάει τέλειωσε. Είμαι αισιόδοξο άνθρωπος οπότε δεν έχουμε κάποια οριστική απάντηση τίποτα δεν έχει χαθεί διότι πραγματικά χρειαζόμαστε την χρηματοδότηση όσον αφορά την εδαφική συνεργασία. Τώρα να επανέλθουμε σε ένα θέμα ε, το οποίο μας απασχόλησε και ας μην είναι τόσο τρομερή νίκη όσον αφορά την απότερη περιφέρεια και εκεί παλέψαμε για να αποσπάσουμε κάποια πράγματα και τα καταφέραμε. Οπότε είπαμε για το ΦΕΝΤΕΡ κάτι να κάνουμε, να κάνουμε το πρόγραμμα BIS. Πρόγραμμα αυτό το οποίο είναι σημαντικό ακόμα και να αφορά ένα μικρό τμήμα της Ένωσης. Επίσης, είναι σημαντικό, όπως είπαμε, να υπάρχει ευελιξία για το 80% όσον αφορά ε, τη, την συγκέντρωση, 80% για αυτά και 20% με ευελιξία, ελεύθερο, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, παλέψαμε για το πώς πάσαμε, επίσης για την πιστοποίηση, για τις ε, ιδιαίτερες προτεραιότητες των προγραμμάτων που έχουν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικά το Back to Interact. Είναι όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε. Ό,τι ζητήσαμε το καταφέραμε. Το πήραμε. Όσον αφορά το ότι δόθηκε και χρηματοδότηση ένα πρόγραμμα, πάρα πολύ σωστό, γιατί έχουν τα κράτη-μέλη θέλουν και υπολογίζουν να ανακτήσουν τους πόρους που έχουν ε, δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα γιατί έτσι είμαστε λιγότερο αποτελεσματικοί. Έχουμε τη σχετική εμπειρία. Πρόκειται κάτι σαν υπόσχεση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δει ότι αναπρόγραμμα τα πράγματα είναι καλύτερα. Επίσης, όσον αφορά το, τη συμπλήρωση των διασυνοριακών προγραμμάτων και εκεί θα συνεχίσουμε με τη βάση της εντολή που υπάρχει, αφού το θέμα δεν έχει κλείσει. Και στο πλαίσιο εντολής, με βάση ψηφοφορία, αποφασίστηκε ποιε είναι οι προτεραιότητες. Ναι, είπαμε, έχετε για την εδαφική συνεργασία παρατηρήσεις, αλλά τέλος πάντων θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Η Μαρίτα Τερέζ μίλησε για τον κανονισμό της εδαφικής συνεργασίας και διασυνοριακή το ΕΟΕΣ για τους ομίλους συμπεριλαμβάνεται και στο κανονισμό για τη διασυνοριακή συνεργασία. Μπορεί να γίνει αναφορά σε αυτό τον κανονισμό λοιπόν. Και κάτι άλλο που καταφέραμε είναι ότι και στα μέσα εξωτερικής πολιτικής γειτονίας και ένταξης οι δυνατότητες ίδρυσης ομίλων προβλέπονται ως ε, μορφές συνεργασίας. Και ευχαριστώ πολύ και του συναδέλφους ε, στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων γι' αυτό. Ο Γιάνν Όλμπριχτ είπε ότι είναι δύσκολο αυτό με τις δημόσιες υπηρεσίες πράγματι και στη Γερμανία λέμε δυο νομικοί τρεις διαφορετικές απόψεις ε, αλλά ε, εμεί είμαστε υπεύθυνοι για το νομοθετικό έργο. Και αν έχουμε τόσο διαφορετικές ε, νομοθεσίες που δεν βοηθάνε να λύνονται τα προβλήματα, τότε θα πρέπει οι νομοθέτες να, και αυτό είναι δική μας δουλειά, θα πρέπει να εργάζονται έτσι ώστε να λύνονται τα προβλήματά με την νομοπαρασκευαστική τους δουλειά. Δεν ότι θα, δεν είπα ότι θα πρέπει να κινηθούν ε, οι νομομαθείς και αυτοί που ορίζουν τον νόμο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά Θα πρέπει κανείς να ορίζει το νόμο στα πλαίσια μιας συνθήκης, άρα δεν είναι απολύτως ελεύθερος να τον ορίσει. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται και για θέμα ερμηνείας των συνθήκων, πρόκειται για μια ε, συνεχιζόμενη διαδικασία. Έχω μια ερώτηση, διότι όταν ε, προετοιμάσαμε τον ε, κανονισμό την πρώτη φορά, μιλήσαμε για τη δυνατότητα για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας να ορίζει όλα τα ευρωπαϊκά ε, προγράμματα. Το ζήτημα είναι κατά πόσο τώρα εντάσσεται στον κανονισμό. Υπάρχει μια διαχειριστική αρχή, ενία διαχειριστική αρχή για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο. Κοιτάξτε πώς έχει το θέμα που το είπαμε στον τελευταίο τριμερή διάλογο. Εδώ δεν είναι εντελώς και νέος κανονισμός, είναι μία τροποποίηση διευρυμένη του υφιστάμενου κανονισμού. Δηλαδή, όλοι οι υφιστάμενοι όμιλοι μπορούν να αποφασίζουν αν θα δουλέψουν με βάση τον παλιό κανονισμό ή αν θα κάνουν χρήση των διευρυμένων δυνατοτήτων του νέου κανονισμού. Και ανάλογα θα προσαρμοστούν Τώρα, οι νεοειδριόμενοι όμιλοι καταρχήν ε, δεσμεύονται από τον τωρινό κανονισμό, αλλά όταν θα επικυρωθεί ο νέος κανονισμός από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που συναποφασίζουν, τότε θα μπορούν να κάνουν χρήση του καινούριου κανονισμού και οι φυστάμενοι όμιλοι μπορούν να προσαρμοστούν, όπως είπαμε, στον ε, νέο κανονισμό. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια δεν υπάρχουν. Ο Νίκολας θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ. Θα πω δύο λόγια κι εγώ. Και θα προσπαθήσω να είμαι θετικός. Αναφέρθηκαν κάποια από αυτά που ήθελα να πω. Εγώ θέλω να εκφράσω για λογαριασμό της Κομισιόν τη μεγάλη εκτίμηση και θαυμασμό του έργου του εισηγητή για όλους τους κανονισμούς ε, των εισηγητών. Ε, είναι μεγάλη δέσμευση που απαιτείται. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, τεχνικά και απαιτούν μεγάλη αφοσίωση. Και αυτό που είδαμε ε, είναι μια προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα, πραγματιστική, ρεαλιστική προσέγγιση, όπου έγινε προσπάθεια να επιτευχθούν ε, οι στόχοι και να επιτελεστεί πρόοδος. Βέβαια, για το, τους, ε, τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις, εκεί δουλεύουμε σε ενότητες. Είναι 18 οι, θεματικές, οι ενότητες. Και τώρα μ, τρεις έχουν κλείσει Οπότε έχουμε συμφωνήσει προσωρινά επί 5 από τις 18 μετά τους 40 τριμερείς διαλόγους. Έχουμε δρόμο να κάνουμε, την επόμενη εβδομάδα ίσως κάνουμε πρόοδο σε 4 ακόμα, οπότε ε, θα έχουμε κάνει τη μισή δουλειά και έχει γίνει ήδη προπαρασκευαστική εργασία για πολλές άλλες ενότητες. Είναι πρόκληση όμως βεβαίως για τους επόμενους τριμερείς διαλόγους, μεγάλες προκλήσεις και η Κομισιόν όπως πάντα θα ε, κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει τη διαδικασία. Γιατί βεβαίως όλοι το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη η σημασία να τηρηθούν οι, τα χρονοδιαγράμματα που ανέφερε η Πρόεδρος και να έχουμε έναν κανονισμό που θα μπορέσει να εγκριθεί τον Οκτώβριο. Είναι κρίσιμο για μας αυτό και αν δεν γίνει δεν θα, έχει μόνο, δεν θα υπάρξουν μόνο πρακτικές συνέπειες για τον προγραμματισμό, αλλά θα είναι αρνητικό και για την γενικότερη πολιτική. Τώρα, για τις τρεις ενότητες που συμφωνήθηκαν και εμείς συμφωνούμε ότι είναι ισορροπημένο το αποτέλεσμα, καλό και εκτιμούμε ως Κομισιόν την υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε ορισμένα κρίσιμα θέματα να διατηρηθούν τα βασικά στοιχεία ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το έργο ελέγχου, της ε, διατάξη για την αναλογικότητα, τις διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων και οικονομικών δημοσιονομικών πληροφοριών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί κρατάει ε, μια ισορροπία σε σχέση με τη συμβολή της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς να αποδυναμώνει άλλες διατάξεις για την επικοινωνία και την πληροφόρηση που είναι σημαντικές. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα, στα οποία, τα οποία χάσαμε και λυπούμεθα γι' αυτό και αφορούν ε, τις 1720 ώρες που ανέφερε η κυρία Κρέλη, η γήτρια. Αλλά αυτό είναι βέβαια κομμάτι της νομοθετικής διαδικασίας. Κάποια στοιχεία δεν θα είναι τέλεια, είναι αναμενόμενο αυτό. Πάντως το αποτέλεσμα είναι καλό. Τώρα, δύο θέματα ετέθησαν σχετικά με τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις. Το performance reserve, το αποθεματικό απόδοση ε, επιδόσεων. Η Κομισιόν ε, ε, το πρότεινε αυτό το αποθεματικό ευθύς εξ αρχή πριν τεθούν θέματα προπολογισμού και το βλέπουμε αυτό ως έναν τρόπο για να δώσουμε ναύσματα για την απόδοση, για τις επιδόσεις. Και μπορεί να εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην δώσει λαβή για τους φόβους που εκφράστηκαν. Και μπορούμε να εξηγήσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα οδηγήσει στις αρνητικές συνέπειες που φοβούνται πολύ και ότι ε, θα έχουμε στις τελικές φάσεις πολλά ε, χρήματα διαθέσιμα. Ε, η τμηματική γενική προσέγγιση έδειξε ότι υπάρχουν διασφαλίσεις, ότι θα υπάρχουν κονδύλια ε, με την προϋπόθεση ότι οι προτεραιότητες ε, δεν θα παρεκκλίνουν και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι θα ε, πείσουμε την διαχειριστική αρχή ότι αν δηλαδή ανταποκριθεί σε σχέση με τις προτεραιότητες τότε θα διατεθούν τα κονδύλια που υπάρχουν. Αυτή λοιπόν είναι μια ιδέα που νομιμοποιείται. Τώρα, για τις, ε, τα ελάχιστα μερίδια, τα, και αυτό είναι κρίσιμο γιατί έχει να κάνει με τη θεματική συγκέντρωση, πρέπει να επιληθεί γιατί επηρεάζει την προγραμματική διαδικασία. Νομίζω από ότι, ε, ε, ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό και είμαστε ανοιχτοί να δούμε διαφορετικούς τρόπους για το πώς θα φτάσουμε στην επίτευξη του τελικού στόχου. Χρειάζεται πιο πολύ δημιουργικότητα για την εξέβρεση λύσεων και εμείς είμαστε ανοιχτοί. Να διερευνήσουμε και άλλες εναλλακτικέ για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας και θα βγούμε από το αδιέξοδο. Ε, τώρα, δύο λόγια για τον κανονισμό του ΕΤΠΑ εδώ χαιρετίζουμε τη στήριξη του Κοινοβουλίου ε, για κάποια βασικά θέματα, ούτως ώστε τα βασικά στοιχεία της θεματικής συγκέντρωσης να παραμείνουν. Είχαμε βέβαια κάποιες επιφυλάξεις για τα νησιά και τη σταδιακή κατάργηση, το phasing out, αλλά οι συμβιβασμοί ε, ε, θέλουν και θυσίες, παραχωρήσεις. Δεν συμφωνούμε ότι η Κομισιόν παγιδεύτηκε ε, σε σχέση με τους θεματικούς στόχους ε, και το, την εξειδίκευση του Ταμείου. Ε, αυτή είναι μια ενιαία προσέγγιση στη χρήση των Ταμείων και ενώ είναι σωστό ότι το ΕΚΤ συμβάλλει σε τέσσερις μόνο θεματικούς στόχους ενώ το ΕΤΠΑ μπορεί δυνητικά σε όλα να συμμετέχει. Κατά τη γνώμη της Κομισιόν δεν θα ήταν χρήσιμο να πούμε ότι κάποιοι στόχοι είναι μόνο για το ΕΚΤ και άλλοι στόχοι είναι μόνο για το ΕΤΠΑ. Και δεν είναι και δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι φτιαγμένα τα ταμεία. Τα κονδύλια του ΕΤΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για το, την κοινωνική ένταξη, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την παιδεία, γιατί υπάρχουν ανάγκες υποδομών που σχετίζονται με αυτά. Είναι η φύση των ταμείων τέτοια που προϋποθέτει μια ενιαία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η δυσκολία, κατά τη γνώμη της Κομισιόν, αφορά τα ελάχιστα μερίδια, η ποσοστά, όταν προσπαθούμε να πάρουμε την θεματική συγκέντρωση που στηρίζεται στα ταμεία, που αφορά όλα τα ταμεία, και να τη συνδυάσουμε με μια συγκέντρωση η οποία ε, στηρίζεται σε θεματικούς στόχους. Εκεί πρέπει να βρούμε μια δημιουργική ε, λύση. Μια συγκεκριμένη ερώτηση αφορούσε την εδαφική συνεργασία και τους ομίλους εδαφικής συνεργασίας. Στον κανονισμό για την εδαφική συνεργασία είναι γραμμένο ότι ένας όμιλος μπορεί να είναι και μια διαχειριστική αρχή. Υπάρχει αυτό στον κανονισμό για την εδαφική συνεργασία και αυτό είναι ένας τρόπος ε, για να προβλέψουμε ότι ε, αυτό το μόρφωμα του ομίλου μπορεί να ε, προχωρήσει τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Μπορεί να είναι διαχειριστική αρχή, μπορεί να είναι ένας δικαιούχος. Και να είναι και δικαιούχο. και στους ομίλους είναι καλό το αποτέλεσμα, είναι πολύ τεχνικός ο κανονισμός, απαιτεί δύσκολες συζητήσεις, αλλά μέσα από την νομοθετική διαδικασία και κρίνοντας εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο ε, εύκολη γινόταν η έγκριση επειδή βελτιωνόταν η πρόταση της Κομισιόν. Και καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα που είναι λειτουργικό και ισορροπημένο επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα θέματα. Τώρα, για το, την εδαφική συνεργασία και το σχετικό κανονισμό, κάτι για τον προϋπολογισμό. Όπως είπε και η Πρόεδρος, είναι πολύ σύνθετο το θέμα λόγω των επιπτώσεων που απορρέουν από τυχόν αλλαγές σε ένα κομμάτι του όλου φακέλου για την πολιτική συνοχή. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της συνεργασίας, όχι μόνο μέσα από τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, αλλά ένας βασικός στόχος, μην το ξεχνάμε, είναι να μην απομονωθεί η εδαφική συνεργασία από την υπόλοιπη πολιτική και θα πρέπει με συμφωνίες να εντάσσουμε παντού το στοιχείο της συνεργασίας και έτσι μπορούμε να ε, συμβάλλουμε σε μακροοικονομικές ε, και μακροπεριφερειακές ε, στρατηγικές λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές της συνεργασίας. Αύριο θα συναντηθούμε με τον Επίτροπο Αλμούνια στις 9 και στην Επιτροπή τώρα γίνονται εσωτερικές διαβουλεύσεις για τις περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές που θα εγκρίνει η Επιτροπή μέχρι τα μέσα Ιουνίου και στις περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές υπήρχε η δυνατότητα να δοθούν ενισχύ στα αεροδρόμια και στον τομέα ενέργειας μέσα στα πλαίσια των περιφερειακών ε, κατευθυντηρίων γραμμών και τώρα η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έχει αποκλείσει αυτούς τους, ε, αυτούς τους δύο τομείς ε, ε, από τις περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό είπε και ο, ο Βίκτορ και σε σχέση με τον τομέα της ενέργειας και για τα αεροδρόμια. Και αυτό αφορά και το Ταμείο Συνοχής, άρα ο αποκλισμός του τομέα της ενέργειας από τις περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή αποκλισμός της ενέργειας από τις περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές, μας οδηγεί σε συμπεράσματα και ως προς τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν ξέρω πώς πρέπει να το ερμηνεύσουμε αυτό, πώς αντιδρά η Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο, πώς το βλέπετε αυτό, αυτό μας ανησυχεί. Θα ρωτήσουμε τον Επίτροπο Αλμούνια αύριο, μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο ή ε, ακολουθείτε την, ε, τη, τη γραμμή της Κομισιόν όπου όλοι έχετε μία και κατευθυντήρια γραμμή. Ναι, αυτό απορρέει από τις συνθήκες. Τι έρχεται πρώτο και τι δεύτερο. Ναι, δεν ξέρουμε, ε, είναι η θεωρία της κότας και του αυγού, ποιος γεννάει ποιον. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι είναι εκλέξιμο ένα αεροδρόμιο το οποίο ε, λαμβάνουμε υπόψη σε επίπεδο συναπόφασης ο Επίτροπος Αλμούνια μπορεί να ακολουθήσει αυτή την υπόδειξη όχι στην ε, πρώην πρόταση του Επιτρόπου Αλμούνια υπήρχε η πρόταση προσθήκης επιπρόσθετων κριτηρίων για τις επενδύσεις που άπτονται το τομέα ενέργειας αλλά τώρα αποκλείονται κομισιόν. Νομίζω ότι ανέκαθεν το θέμα την σχέση μεταξύ των περιφερειακών κατευθυντηρίων και των κεντρικών. Επομένως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια διάρθρωση που πρέπει να γίνει, η συνάρθρωση για αυτές τις ε, κατευθυντηρίες που αναφέρονται στο ότι ορισμένες προϋποθέσεις που προέρχονται από τις κεντρικές θα πρέπει να πληρώνται. Όσον αφορά την ενέργεια, η τρέχουσα θέση σε σχέση τι προτείνεται είναι το ότι εν προκειμένου το θέμα της κρατικής βοήθειας αφορά τις καθεντηρίες. Γιατί ακόμα δεν έχουμε μια πλήρη εμφάνιση παρουσίαση προβολή τους. Να δούμε τι ισχύει σχέση με ό,τι προβλέπουμε. Εκτός μικροφώνου η πρόεδρος για τις τομεακές κατευθυντήριες. Να δούμε κατά πόσον αυτό βοηθάει τις ε, επενδύσεις μας. Θα το δούμε αυτό αύριο. Κομισιόν. Ο κύριος Αλμούνιο μόνο μπορεί να σας πει. Δηλαδή η Γενική Διεύθυνση του Ανταγωνισμού. Πάντως για το γενικότερο θέμα το οποίο έδειξε ο κύριος ε, Όμπρεκτ. Ε, ο κανονισμός των κοινών διατάξεων λέει τι ισχύει όσον αφορά τις επενδύσει της πολιτικής συνοχή. δυνάμει των κανόνων που διέπουν τι κρατικέ ενισχύσει. Οπότε, εξ όλα, θα πρέπει όλα αυτά να συνάδουν προ τι διατάξει που διέπουν τις κρατικέ ενισχύσει. Βεβαίω, όσον αφορά τη διαμόρφωση του τοπίου για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνέχεια με τους στόχους της πολιτικής, αλλιώς δεν έχει νόημα. πολιτική δηλαδή των επενδύσεων, πολιτική συνοχή. Να δούμε δηλαδή, λόγω των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, ποιες επενδύσεις ε, ωφελούνται και ευνοούνται. Βέβαια, δεν θα θεωρήσουμε ότι δεν συνάδει και αντιφάσκει. Αν έχουμε κάποιους περιορισμούς που αφορούν τους, τους κανόνες των ενισχύσεων όσον αφορά την ε, ένταση της ενίσχυσης, τις ε, προϋποθέσεις που αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, τέλος πάντων κάποια επιπλέον στοιχεία σε σχέση με τους πόρους του Ταμείου Συνοχής ή της πολιτικής συνοχής. Απλώ κάθε φορά πρέπει να εξετάζονται οι στόχοι κάθε πολιτικής Όλμπριχτ. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αλλά να μην ξεχάσουμε προς τα πού πάμε, σε τι σκοπός υπάρχει, τι είναι επιλέξιμο κάθε φορά και τι απαγορεύεται. Είναι θέμα κοινωτικού δικαίου. Εμείς επεξεργαζόμαστε έναν κανονισμό και κανονίζει για Στις κρατικές λένε ότι κάτι δεν ισχύει το οποίο εμείς το σβήνουμε μετά τον κανονισμό. Τι λέτε, έτσι είναι, κομισιόν. Ναι, θα πρέπει κάποιος να προσέξει όταν μιλάει για επιλεξιμότητα. Γιατί δεν αποκλείεται, επί τη βάση του κειμένου, δεν αποκλείεται να προβλέπεται ενίσχυση, υποστήριξη, βοήθεια προς αεροδρόμια. Σε σχέση επίσης και με την προστασία του περιβάλλοντος όταν έχουμε ας πούμε επένδυση από κάποια εταιρεία η οποία ενεργώντας παραβλάπτει το περιβάλλον. Κάπως έτσι το βλέπω. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Όλμπριχτ. Κομισιόν, να το δείτε. Ευρύτερα, πέρα από την περιφερειακή ενίσχυση. Γιατί ακόμα και αν έχουμε ακόμα και αν επιτρέπουν οι κανόνες τη περιφερειακή πολιτική μια ε, ρύθμιση, τότε μπορεί να απαγορεύεται από αλλού. Τόσο το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Τα κρατημέλη μπορούν να έχουν την επιλογή τι είδου ενίσχυση θέλουν να επικαλεστούν κάθε φορά και να κάνουν την κοινοποίηση για να μπορέσουν να πάρουν την έγκριση για να χορηγηθεί η κρατική ενίσχυση. Παρακαλώ αύριο οι ενισχυτές να ξεκαθαρίζουν αυτά τα θέματα. Μπορώ, μπορείτε να το κάνετε ρωτώντα τον Επίτροπο Αλμούνια. Άρα να κλείσουμε αυτό το θέμα. Το κλείσαμε, το ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκολα τη Επιτροπή. Ε, ε, if... Και θα κάνουμε τη συνεδρίαση τώρα των συντονιστών. Φωνάξτε τους συντονιστές σας γιατί αλλιώς θα αποφασίσουν και θα είναι εδώ, γιατί θα είναι εδώ, μόνο η, η ECR, το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές. Άρα σε λίγα για να έρθουν όλοι εδώ. <laughs>